Αγαπητοί συνάδελφοι, σας ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά μετά το χθεσινό τριμερή διάλογο για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο είχα κάποιες επίγουσες συνομιλίες σήμερα με μία μικρή καθυστέρηση για την οποία ζητώ συγγνώμη και από τους διερμηνείς αλλά και από όλα τα μέλη της Επιτροπής. Περνάμε στο σημείο 17 και δίνω το λόγο στην συνάδελφο Καρή Μαντελή για να μας παρουσιάσει τις 326 τροπολογίες που κατατέθηκαν επί της έκθεσης πρωτοβουλίας της με θέμα την κοινωνική στέγαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση να σας ε, επισημάνω επίσης ότι σε λίγο θα έρθει, φαντάζομαι θα έχει και εκείνος κάποια τηλεφωνήματα να κάνει, ο Ρέιμον Χάνκ που είναι εισηγητής για το ίδιο θέμα στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Αν έρθει λοιπόν, πολύ ευχαρίστω να δώσω το λόγο. Προς το παρόν όμως ακούσουμε τη δική μας εισηγήτρια, την κυρία Καρή Μαντελή. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τους σκιώδεις ηγητές μας για την συμβολή τους και όλους όσους συνέβαλαν στον εμπλουτισμό της έκθεσης. Θα ήθελα να επισημάνω ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα που έχουμε στο κοινοβουλευτικό έργο, γιατί αναχαιτίστηκε κάπως το έργο μας εξαιτίας ε, κάποιων προβλημάτων ε, στη μετάφραση μεταξύ γαλλικής και αγγλικής ε, εκδοχής. Αυτό και ως προς την έκθεση και ως προς τις τροπολογίες. Χρειάστηκε λοιπόν να καταθέσω πολλές ε, ε, γλωσσικές τροπολογίες για διορθώσεις των μεταφράσεων. Η έκθεση αυτή λαμβάνει υπόψη, αγαπητοί συνάδελφοι, την ανησυχητική κατάσταση σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στη στέγαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί η κοινωνική και οικονομική κρίση διακυβεύει ένα θεμελιώδης δικαίωμα, το δικαίωμα πρόσβαση στην κατοικία. Και παντού σήμερα στην Ευρώπη πολλοί, πολλά νοικοκυριά, πολλοί Ευρωπαίοι συμπολίτες μας δεν έχουν ε, τα μέσα, τα, τους πόρους να αγοράσουν μια αξιοπρεπή κατοικία εξαιτία της αύξησης ε, και των νοικίων και των δημών ενέργειας. Γι' αυτό και η διέκθεσή μας ε, είναι πολύ σημαντική, γιατί η κοινωνική στέγαση ε, μπορεί πραγματικά να αποσβέσει τους οικονομικούς και κοινωνικούς κραδασμούς. Γι' αυτό και η έκθεσή μας ε, ε, καλεί σε ουσιαστικές επενδύσεις στον τομέα αυτό για να καλύψουμε τις κατεπίγουσες κοινωνικές ανάγκες και να ανταποκριθούμε στις ανάγκες των συμπολιτών μας που δυστυχώς σήμερα διαβιούν σε συνθήκες άθλιες. Γι' αυτό με την έκθεση ε, καλούμε ε, για επενδύσεις στον τομέα αυτό της κοινωνικής στέγασης και εξάρουμε το ρόλο της κοινωνικής στέγασης ως ε, οικονομικού σταθεροποιητή. Αυτό πολύ συχνά το ξεχνάμε, αλλά η κοινωνική στέγαση σήμερα είναι σημαντική, γιατί όσο περισσότερες κοινωνικές κατοικίες έχουμε σε ένα κράτος, τόσο πιο εύκολα θα αναχαιτήσουμε το φαινόμενο της ε, φούσκας των ακινήτων. Ο κατασκευαστικός τομέας που σήμερα δυστυχώς βρίσκεται σε ύφεση εξαιτίας της κρίσης είναι ένας κλάδος που θα επιτρέψει μια αύξηση των ε, τοπικών θέσεων απασχόλησης και θα μπορέσει μια νέα άθηση του οικοδομικού κλάδου να αποτελέσει κινητήριο μοχλό και ολόκληρης της ε, οικονομικής ανάκαμψης. Βρισκόμαστε στα πρόθυρα μια σημαντικής ε, μεταρρύθμισης ε, και μεταμόρφωσης και ενεργειακής και θα μπορέσουμε ταυτόχρονα να αναπτύξουμε την πράσινη οικονομία, την τοπική οικονομία και να προσαρμόσουμε τον τομέα, λαμβάνοντας υπόψη και την ανάγκη της κατάρτισης. Η με μεταρρυθμίσει αυτέ θα πρέπει να είναι δικέ και στην, στο θέμα τη στέγασης. Και επίση να αντιμετωπίσουμε και το θέμα του επισφαλού χαρακτήρα τη ενέργεια. Έχουμε μια νέα πρόκληση σήμερα με πολύ σοβαρέ συνέπειε στο βιωτικό επίπεδο και στα ποιότητα ζωή των συμπολιτών μα Και η έκθεση το επισημαίνει αυτό. Επί τη ουσία τώρα θα ήθελα να σα αναφέρω δύο-τρία σημεία για τα οποία ζητώ και την υποστήριξή σας. Καταρχήν ε, θα θέλαμε να ιδρύσουμε ένα ευρωπαϊκό παρατηρητήριο στέγασης ε, για να συλλέξουμε εθνικά στατιστικά στοιχεία, να ενθαρρύνουμε την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και να συνδράμουμε τα κράτη-μέλη ώστε να μπορέσουν να διαμορφώσουν την πολιτική στέγασης, ε, ιδιαίτερα λαμβάνοντα υπόψη την ανάγκη κοινωνική στέγαση και μια πολιτική για τι προσιτέ τιμέ τη κατοικία. παράγραφος 5. Δεύτερη ε, σημαντική ιδέα. Στα πλαίσια τη οικονομική διακυβέρνηση και του ευρωπαϊκού εξαμήνου να δημιουργήσουμε ένα πίνακα κοινωνικών δικτών, Όπω επενδύσει στην κοινωνική στέγαση. Θέλουμε να αποτιμήσουμε τις πρόοδου το κρατών στον τομέα αυτό. Τροπολογία 111. Επίση, να δημιουργήσουμε ένα μηχανισμό ε, στα κράτη-μέλη για την περίοδο της ύφεσης των ισχυρών Αγιολάδων και επίσης ε, είχαμε ένα σχετικό, ε, μια σχετική έκθεση για τους αστέγους που την εγκρίναμε και με συντριπτική πλειοψηφία. Για να αποφύγουμε λοιπόν την έξαρση του φαινομένου των αστέγων ε, θα πρέπει να τους κρατήσουμε στα σπίτια τους και νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό αυτή της χειμερινής εκεχηρίας κατά κάποιο τρόπο αυτή η πρόταση συνεργάστηκα με τους ε, σκιώδεις ηγητές ε, και προσπάθησα να συμπηλήσω τις ε, τροπολογίες σε μερικές συμβιβαστικές τροπολογίες που μοιράστηκαν χθε το βράδυ και ευελπιστώ ότι με την έκθεση αυτή θα μπορέσει και η Επιτροπή μας να επηρεάσει άμεσα την καθημερινότητα των συμπολιτών μας. Γιατί μιλούμε για κοινωνική στέγαση, το πιο θεμελιώδες δικαίωμα και θεωρώ, ευελπιστώ μάλλον, θα καταλήξουμε σε πολύ καλές συμβαστικές τροπολογίες για να υπερψηφίσουμε την έκθεση. Σας ευχαριστώ. Ο Αλεχάνδρο Σέρκας και μετά ο Φιλίπ Μπένιον. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω πρώτα απ' όλα ότι το θέμα της κοινωνικής στέγασης ε, είναι κάτι που για την ομάδα μου αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα, ιδιαίτερα στους χαλεπούς καιρούς της κρίσης, όπου πολλοί συμπολίτε μας όχι μόνο έχουν πρόβλημα στην πρόσβαση της, στην κατοικία, αλλά και εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι εξαιτία της κρίσης και της ανεργίας ε, χάνουν την κατοικία τους, υπόκειται σε έξωση και αντιμετωπίζουν τεράστιες κοινωνικές αδικίες. Η Καρή Μαντελή με πολύ εύστοχο και προοδευτικό τρόπο συνέταξε την έκθεσή της. Εμείς ε, καταθέσαμε 39 τροπολογίες και θα ήθελα να σας περιγράψω τις πιο σημαντικές που περιστρέφονται γύρω από τρεις άξονες που είναι σημαντικοί για τους σοσιαλιστές και εκεί θέλουμε να εμπλουτίσουμε και να βελτιώσουμε την έκθεση Καρή Μαντελή. Θεωρούμε ότι θα πρέπει καταρχήν να, ε, να εξάρουμε την ε, ανάγκη μιας ευρωπαϊκής πολιτικής, γιατί στην έκθεση πρωτοβουλίας δεν υπάρχει κάτι τέτοιο ξεχωριστό. Θα θέλαμε ένα τίτλο πραγματικά για την ευρωπαϊκή πολιτική. Όχι μόνο συστάσεις ε, προς τα κράτη-μέλη, τι πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κοινοτικά θεσμικά όργανα, η Επιτροπή, το Κοινοβούλιο. Και από την άποψη αυτή να υπενθυμίσουμε το άρθρο 14 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το πρωτόκολλο 16. Δεν είναι κάτι που ε, επινοούμε σήμερα αν υπήρχαν προηγουμένω νομικέ βάσεις για τέτοια πολιτική. Μίλησε για την ανάγκη δικτών στο ευρωπαϊκό εξάμεινο. Το ζητούμε και εμείς με τις τροπολογίες και επίση θέλουμε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο ένα πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση που να εξασφαλίζει μια συνεκτικότητα των κοινοτικών πολιτικών που έχουν επίδραση στην κατοικία και που είναι κάπως δεσπαρμένες, κατασπαρμένες όπως ε, το θέμα της ευημερίας, των διαθετικών ταμείων, ενέργεια, υγεία, καταπολέμηση της ε, φτώχειας και της ε, ανισότητας. Πρόκειται για κοινοτικές πολιτικές που υπό διαφορετικές σκοπιές και πρίσματα επηρεάζουν την πολιτική της στέγασης και της κατοικίας, αλλά δεν υπάρχει μία ενιαία συντονισμένη στρατηγική και την ανάγκη αυτής της πολιτικής επισημαίνουμε. Επίσης, έχουμε την πολιτική ανταγωνισμού. Η πολιτική ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης όχι μόνο δεν εξυπηρετεί τους στόχους της Ευρώπης ε, του 2020 και την καταπολέμηση των ανισοτήτων ε, ή το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, αντίθετα ε, αντιβαίνει, αντιμάχεται αυτή, αυτούς τους στόχους. Και μάλιστα όταν ε, έχουμε μία αντιπαράθεση της πολιτικής ανταγωνισμού και της πολιτικής αγοράς με την κοινωνική πολιτική, ουσιαστικά το θύμα αυτής της ε, αντιπαλότητας είναι η κοινωνική στέγαση στα κράτη-μέλη. Το είδαμε στη Σουηδία, στην Ολλανδία, στην ε, Γαλλία. Θα πρέπει λοιπόν να επανεξετάσουμε αυτή την πολιτική του ανταγωνισμού για να την ευθυγραμμίσουμε και να τη συντονίσουμε με τις κοινωνικές πολιτικές. Αυτό ζητούμε στην πολιτική 16, να διευκρινιστούν οι στόχοι της πολιτικής ανταγωνισμού για να αποφευθούν οι αντιφάσεις. Επίσης, να συνδυαστεί με την πολιτική, τη στρατηγική για το 2020 και να γίνουν σεβαστές οι αρχές υπέρ των κοινοφελών υπηρεσιών. Και στην τροπολογία 21 ζητούμε αναθεώρηση του πακέτου για τις κρατικές ενισχύσεις του 2011, που όχι μόνο δεν ε, επιλύει τα προβλήματα της κοινωνικής στέγασης, αλλά εμποδίζει τα κρατημέλη να συνεχίσουν τις αυτόνομες πολιτικές τους και παρόλο που κάποια κρατημέλη δεκαετίε δεκαετίες ολόκληρες είχαν εφαρμόσει δίκαιη και αποτελεσματική λύση, τα, εμποδίζουμε, εμποδίζουμε να τη συνεχίσουν. Επίσης, ε, θα πρέπει να σταματήσουμε ε, μια νομοθεσία και νομοθετικέ διατάξει ε, για τα ενυπόθηκα δάνεια που ουσιαστικά εξουδετερώνουν τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών. Έχουμε ε, την τροπολογία 10. Αυτά, αυτές οι, αυτοί οι κανόνες για τα ανυπόθηκα δάνεια εξυπηρετούν μόνο το τραπεζικό σύστημα και α, ταλανίζουν τους πολίτες, γιατί οι τράπεζες δεν αναλαμβάνουν κανένα απολύτως κίνδυνο, ενώ τα νοικοκυριά, οι οικογένειες, οι συμπολίτες μας εξωθούνται σε οικονομική εξαθλίωση και σε χρεοκοπία οι άνθρωποι χάνουν τα σπίτια τους ε, στην Ισπανία και παρόλα αυτά συνεχίζουν να είναι υπόχρεοι απέναντι στις τράπεζες για να εξυπηρετήσουν τα δάνειά τους. Οι τράπεζες μόνο για το κέρδος ενδιαφέρονται, ενώ οι άνθρωποι χρειάζεται να καταβάλουν ε, τοκογλυφικά δάνεια και μερικές φορές ε, λόγω αδυναμίας αποπληρωμής χάνουν το σπίτι τους, αλλά η ευθύνη, η νομική υποχρέωσή τους να αποπληρώσουν το δάνειο συνεχίζεται. Είναι παράλογο αυτό, είναι μια τραγωδία στην Ισπανία. Είχαμε ευτυχώς μια απόφαση 415 που ε, ουσιαστικά απαξιώνει αυτή την νομοθεσία. Αλλά το θέμα είναι να μην σταματήσουμε στις δικαστικές αποφάσεις. Θα πρέπει και οι νομοθέτες να αναθεωρήσουν αυτή τη διαδικασία για τα ενυπόθηκα δάνεια, ώστε να στραφεί το πρίσμα από την εξυπηρέτηση των τραπεζών στην εξυπηρέτηση των συμπολιτών μας. Θα πρέπει και οι τράπεζες να αναλαμβάνουν τον κίνδυνο. Και μια και οι επιχειρήσεις έχουν δυνατότητα στα πλαίσια της ε, χρεοκοπίας σε διάφορες ε, ε, θετικές διατάξεις, θα πρέπει τα ίδια πλονεκτήματα που δίνουμε στις επιχειρήσεις σε περίπτωση χρεοκοπίας να τα χορηγήσουμε και στους συμπολίτε μας, για να έχουν και μια δεύτερη ευκαιρία, όπως έχουν συνήθως και οι έμποροι όταν χρεοκοπούν. Θέλουμε λοιπόν μια ισχυρή έκθεση να διατρανώσουμε την ευρωπαϊκή άποψη για να καταλάβουν οι πολίτες ότι ενδιαφερόμαστε για αυτούς. Θα δώσω το λόγο στον Φιλίπ Μπενιόν τώρα, αλλά δεν αντιστέκομαι σε ένα σχόλιο σε ό,τι αφορά το αίτημα για κοινοτική νομοθεσία ως προς τα ενεπόθηκα δάνεια. Είναι παλιό το θέμα και μάλιστα είναι κάτι που το διεκδικεί πια και ο τραπεζικό τομέα, γιατί έτσι θεωρεί ότι ε, θα διευρυνθεί η δυνατότητα προσφορά ενυπόθηκων δανείων. Θα πρέπει λοιπόν να θεσπίσουμε νομοθεσία για τα ενυπόθηκα δάνεια, αλλά ε, να εξασφαλίσουμε πρώτα απ' όλα τα δικαιώματα των χρηστών, των ε, συμπολιτών μας, των πολιτών και όχι να δώσουμε νέες ευκαιρίες στους στη δημιουργικότητα και την καινοτομία των τραπεζιτών. Ο Φιλίπ Μπενιό. Uh, thank you. very much like to thank the Θα ήθελα να ε, ευχαριστήσω την συγγήτρια, διότι πραγματικά γίνεται μια αξιοπρεπέστατη προσπάθεια για να σημειωθεί επιτέλους πρόεδρος ε, σε αυτό το θέμα και είναι κοινή προσπάθεια όλων πριν από την σύνταξη της έκθεσης είναι ένα σεμινάριο χάρη στο οποίο όλοι μεταξύ των οποίων και εγώ ε, προσφέραμε μια συνδρομή και καταθέσαμε τροπολογίες. Δεν χρειάζεται τώρα να τις διατρέξουμε όλες γιατί είναι πάνω από 300 και στις 10 ακόμη αυτό θα συζητάμε αλλά για θεματικές ενότητες διάφορες τροπολογίες αποσκοπούν στην προσθήκη του όρου affordable, σε προσιτή τιμή. Διότι στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε έναν τεχνικό ορισμό που αντικατέστησε τον όρο κοινωνική στέγη, διότι ε, δεν είναι μονοκρατικό το ζήτημα. Υπάρχουν ε, φορεί κρατική, αλλά και ιδιωτικοί που παρέχουν την κοινωνική στέγη. Στη συνέχεια, όπω σα έλεγα, υπάρχουν ε, διάφορε τροπολογίε για να αναφέρεται τη συμμετοχή και του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Επίση, θα ήθελα κάποιε διευκρινήσει μέσα από τι τροπολογίε μου για τι κρατικέ επιδοτήσει. Χρειάζεται μία ισορροπία ανάμεσα ε, στη συμμετοχή του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, κυρίως όταν μιλάμε για κρατικέ επιδοτήσεις και τους σχετικούς κανόνες. Mm. Προσιτή τιμή, λοιπόν, πρέπει να λάβουμε υπόψη το κόστος των τιμολογίων για τη θέρμανση κυρίως, ούτως ώστε η κοινωνική στέγη αλλά και η ιδιωτική στέγη ε, θα είναι σε προσιτή τιμή χάρη σε μέτρα ενεργειακής αποδοτικότητας. Ε, θα πρέπει να μπούμε σε έναν ενάρετο κύκλο χρησιμοποιώντας ένα συνδυασμό εθνικής ε, και ενωσιακής χρηματοδότησης εισερχόμενη σας λέω σε έναν ενάρετο κύκλο και αποκτώντας μια μόχλευση αξιοποιώντας ε, έτσι τα ωφέλη με ε, τρόπο ώστε να χρηματοδοτήσουμε και μελλοντικά προγράμματα. Επίσης θα χρειαστεί να επικρατήσει σαφήνεια ως προς τις εθνικές και ενωσιακές αρμοδιότητες. Ε, είμαι πεπισμένος ότι θα καταλήξουμε σε ικανοποιητικές συμβαστικές λύσεις και προσβλέπω στο επόμενο στάδιο των διαβουλεύσεων μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ιζαμπέλ Μογάν Σαχτιέλη, πρόεδρος, Αν Σανκλέρ, στη συνέχεια ε, θα ήθελα να μάθω αν ζητήσει κάποιος άλλος το λόγο μετά από τους, τα δύο αυτά μέλη εντάξει, άρχισα με ελαφρία καθυστέρηση, ζήτησα συγγνώμη, τι να κάνω, έχουμε αργοπορήσει ε, και θα καθυστερήσει και είναι των, ε, της ψηφοφορίας ως τι να κάνουμε. να κλείσω τον κατάλογο των ομιλητών. Ο κύριος Ρέιμουρ Χάγκη, Α, όχι, δεν ζητάει τον λόγο. Ένα λεπτά και εκπρόσωπο Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπάρχει και δεν. Α, ούτε. Καταπληκτικό. Μωράν Σαρτιέ, Σανκλέρ, η συγγήτριά μα μετά. Και θα περάσουμε στο επόμενο σημείο. Μα θα είμαι πολύ σύντομη, Πρόεδρε. Δεν χρειάζεται να χειροτερέψω και εγώ την καθυστέρηση που έχουμε ήδη. Ευχαριστώ την κυρία Ντελή που ασχολείται πισταμένα με αυτό το ζήτημα. Δίκαιο έχει. Ε, ενώ αγωνιζόμαστε τώρα στα πλαίσια του τριμερούς διαλόγου για να ε, σώσουμε το κομμάτι του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ε, και τα κονδύλια που διοχετεύονται ε, στην καταπολέμηση της ένδυας, θα την ενθαρρύνω. Ε, ε, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, μεταξύ άλλων, έχει και αυτό το στόχο καταπολέμηση στόχια μέσω τη κοινωνική στέγη, μεταξύ άλλων. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε ένα ευρωπαϊκό όραμα για την κοινωνική στέγη. Τα δύο αυτά τα ζητήματα είναι αλληλένδετα και ε, χρειαζόμαστε την έκθεση της κυρίας Καρή Μαντελή για να υποστηριχθεί η εργασία που κάνουμε για να σώσουμε αυτά τα κονδύλια του ΕΚΤ. Έχω καταθέσει διάφορες τροπολογίες με στόχο την αναβάθμιση της ενεργειακής αποδοτικότητας ε, στην κοινωνική στέγη. Συνειδητοποιούμε ότι στους ε, φτωχότερους, στα φτωχότερα νοικοκυριά, ε, η προσπάθεια του ελέγχου της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτηρίων ε, λάβει δια της απουσίας της και την ευχαριστώ την εισηγήτρια που τα έλαβε όντως υπόψη στην έκθεσή της. Ευχαριστούμε κυρία Σινκλέρ. Ευχαριστώ. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η κοινωνική κατοικία είναι σημαντικό κομμάτι των ε, κοινωνιών μας. Αυτό αφορά και εμένα βέβαια, γιατί και εγώ ξέρετε σε τέτοιου είδου ε, κοινωνική κατοικία μεγάλωσα. Βεβαίως ε, τα τελευταία 18 χρόνια ε, δεν υπήρχε χρηματοδότηση και με την τελευταία εργατική κυβέρνηση ε, μόνο 14.000 άνθρωποι είχε υποθεί ότι θα έρθουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό βέβαια ήταν ένα βάρος ε, για την ε, κοινωνική τοπική αυτοδιοίκηση. Όπως ξέρουμε τελικά δεν ήταν 14.000 αλλά περίπου ένα εκατομμύριο. Και του χρόνου από ό,τι φαίνεται θα έρθουν και άλλοι από την Ανατολική Ευρώπη και η κυβέρνηση συνασπισμού εξακολουθεί να μην μας λέει πόσοι θα έρθουν. Ε, το θέμα είναι η τοπική αυτοδιοίκηση πώς θα προγραμματίσει την κοινωνική κατοικία. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, μεγάλο βάρος ε, στην ε, τοπική κοινωνία τουλάχιστον για την ε, δική μου την ε, περιφέρεια. Ε, δεν μπορούν βέβαια να τους αρνηθούν, όμως μερικοί αρνήθηκαν γιατί δεν τους άρεσε η κουζίνα. Ήθελαν να τους εγκαταστήσουν μια νέα σύγχρονη κουζίνα. Μήπως οι άνθρωποι αυτοί έχουν ιδιαίτερα δικαιώματα. Σας ευχαριστούμε η Σας ευχαριστούμε Τώρα. Chers euh, ε, αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις και τις τροπολογίες σας. Ε, δεν νομίζω ότι συνιστά πρόβλημα η κοινωνική στέγη. Λύση είναι για τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από την κρίση της στέγης που βιώνουμε σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ε, θα προσπαθήσω να καταλήξουμε στις συμβαστικές τροπολογίες, αλλά ο αγώνας ε, δεν σταματά στο Κοινοβούλιο, το ίδιο θα συμβεί και στην Επιτροπή και στα κράτη-μέλη, ούτως ώστε όλοι να ε, ασκήσουν το θεμελιώδες δικαίωμά τους στη στέγη. Ως προς την ενεργειακή αποδοτικότητα και την ενεργειακή επισφάλεια είναι ένα κεντρικό κομμάτι της έκθεσής μου Γι' αυτό το λόγο ενισχύουμε τις επενδύσεις σε αυτόν τον τρόπο. σας έλεγα στην παρουσίασή μου. Αυτό επηρεάζει άμεσα και την ανεργία, διότι Πρόκειται για θέσεις απασχόληση σε πράσινου τομεί τη οικονομία, νέου τομεί της οικονομίας που μελλοντικά θα γνωρίσουν σημαντική ανάπτυξη. Είπα και μία νοησία προηγουμένω. Ε, σα είπα ότι οι συμβαστικέ τροπολογίε ε, θα σα σας έχουν ήδη σταλεί. Δεν σας έχουν σταλεί σήμερα το βράδυ. Θα σας τη στείλω και την επόμενη εβδομάδα θα καλέσω τους Κιώδης και είμαι σίγουρη ότι θα έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα. Πρόεδρο, σας ευχαριστούμε. Θα εξετάσουμε τις συμβαστικές τροπολογίες, οποίες μόλις αναφερθήκατε στις 22 Απριλίου. Ε, την ΕΠΑΒΡΙΟ 23 θα ψηφίσουμε. Ολοκληρώνουμε το σημείο αυτό της μέσης διάταξης και θα αρχίσει η ψηφοφορία. Σημείο 18 πρώτα απ' όλα. Θα ψηφίσουμε την επιστολή που προετοίμασε η ομάδα εργασία τη Επιτροπή Απασχόληση για Ταμείο Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση. Μια, ε, μια Αυστριακή ε, περίπτωση στην καπνοβιομηχανία. Στην Αυστρία η καπνοβιομηχανία έπεσε θύμα ενός διπλού φαινομένου παγκοσμιοποίησης ως προς την κατανάλωση αλλά και ως προς την παραγωγή μειώνεται η κατανάλωση, ενώ αυξάνεται ε, στην ε, Κίνα, στη Ρωσία και σε άλλες χώρες που τώρα ανακαλύπτουν τα θέλη της καταναλωτικής μας κοινωνίας και υπάρχει και το πρόβλημα στην τομέα της παραγωγής. Σε ποιήν υπέρ, κατά... Α, θα κάνουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία. Έναρξη, έχετε τις κάρτες σας μαζί.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 Εγκρίνεται. Δεύτερο, για την Επιτροπή Προπολογισμών Λαμασούρ για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση στην περίπτωση μια ε, ε, επιχείρηση ε, αζίλ ονομάζεται στην Ιταλία Ε, εταιρεία ε, τεχνολογιών ε, επικοινωνίας και πληροφορικής με έντονη παρουσία σε όλη την Ιταλική επικράτεια. Παρακαλώ ψηφίζουμε. Πέρας. υπέρ, 3 ψήφικα κατά, μηδέν αποχές, εγκρίνεται η επιστολή. Nous en venons τώρα 20. Φτάσαμε τώρα στο σημείο 20. Θα ψηφίσουμε για τη γνωμοδότηση του συναδέλφου Τσάμπα Σόγκορ με θέμα την ε, την εκπαιδευτική και επαγγελματική κινητικότητα των γυναικών στην Ευρώπη. Γνωμοδότηση με αποδέκτη την Επιτροπή Γυναικών, όπου η συγγήτρια είναι η Λουτσία Ουζολή, συνάδελφό μα. Ε, πρώτη τροπολογία τη κυρία Μπλίνκεβίτσετα. Υπέρ, κατά αποχέ εγκρίνεται. τα συμβαστική Β από τέσσερι ομάδε υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά, τροπολογία 3, Μπλίνκεβιτς ούτε υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 4, της υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 2, 7, Τσούμπερ, υπέρ, κατά, αποχές, Νομίζω απορρίπτεται, αλλά θα γίνει επαλήθευση με ηλεκτρονική ψηφοφορία, έναρξη. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Ψήφισαν όλοι. Έβαλαν όλοι τις κάρτες τους. Όλα καλά. Πέρας. 23 ε, υπέρ, 19 κατά, 0 αποχές. Εγκρίνεται η τροπολογία 7 της κυρίας Τσούμπερ, αντίθετα με αυτό που πίστευα. 6 Μπλίνκεβιτσούτ ε, υπέρ, κατά. Θα κάνουμε την εξακρίβωση. Νομίζω ίδιο θα είναι το αποτέλεσμα. Μία επαλήθευση για την 6 παρακαλώ ψηφίστε. Πέρας. 24 υπέρ, 19 κατά. Όντως, εγκρίθηκε. Η τροπολογία 5, King Kings, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Μετά, τροπολογία 8, Τσούμπερ, υπέρ, κατά, αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται επαλήθευση για την 8 της κυρίας Τσούμπερ. Πέρας. 19 υπέρ, 23 κατά αυτή τη φορά καταψηφίστηκε. Ε, τέσσερις πολιτικές ομάδες, συμβαστική α υπέρ κατά ε, αποχές εγκρίνεται. Στη συνέχεια 10 κορνέλισεν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά 11 Μπλίνκεβιτσούτε και προφορική τροπολογία. Δεν υπάρχει ένσταση για την προφορική τροπολογία. Θα ψηφιστεί έτσι η 11 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 2.12 12 τσούμπερ υπέρ, κατά αποχές επαλήθευση. Ηλεκτρονική ψηφοφορία για τη 12. Άρχεται. Ψήφισαν όλοι πέρες. 27 υπέρ. 12 κατά. Ξεκάθαρε υπερψηφίστηκε. 13 εν υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 14 Μπλίκεβιτσούτε υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 18 εν υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 19 εν υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 4, συμβαστική δέλτα, 4 πολιτικές ομάδες υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 5, 21, Κορνέλης, εν υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 22, Μπλίνκεβιτσούτε, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 6, 23, Σόγκορ, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 7, ε, συμβαστική σε τεσσάρων πολιτικών ομάδων υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται μετά την παράγραφο 7, 26 εσάια υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 27 κορνέλης εν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται μετά την παράγραφο 8 συμβαστική ε, ε 4 πολιτικών ομάδων υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, παράγραφος 8, ε, το δεύτερο εδάφιο, τροπολογία 32 Πλικεβιτσούτε, προφορική τροπολογία δεν υπάρχει ένσταση, ψηφίστε για την 32 όσο έχει, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, η 30 Κίνκα Γκιόνσε είναι συμβατή, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 33 Μπλικεβιτσούτε, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 34 εν υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 36 Τσούμπερ υπέρ. Κατά αποχές επαλήθευση. Τσούμπερ 36 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Άρχεται. Πέρας. 19 υπέρ, 16 κατά. Εγκρίνεται. Παράγραφος 10, 37, Κορνέλησεν υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 38 Μπλικεβίτσου είναι συμβατή. Ψηφίζουμε με προφορική τροπολογία. Δεν υπάρχει ένσταση για την προφορική. Ψηφίζουμε ως έχει υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 12, 39, σόγκορ υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 12, 40 της Κορνέλησεν, ναι, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 12, τροπολογία 41, Μπλικεβιτσιούτεν, προφορική τροπολογία υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 42 ε, με τις, ε, της ιδίας, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Θα ψηφίσουμε για το σύνολο της γνωμοδότησης με ηλεκτρονική ψηφοφορία, παρακαλώ. Ε, Πήγε ψήφισαν όλοι. Ε, πέρασε ψηφοφορίας. 40 ψήφοι υπέρ, 3 κατά, καμία αποχή. Συγχαρητήρια στην εισηγήτριά μας. Et nous en venons au point. Περνάμε στο 21. Στην αγνομαδότηση της κυρίας Μακιντάιρ προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Πρόκειται για έκθεση με βάση την οδηγία του Συμβουλίου ως προς, βασικές, ως προς βασικούς κανόνες ασφαλείας για την υγειονομική προστασία από τους κινδύνους που προκύπτουν από την έκθεση σε ιονίζουσες ακτινοβολίες, για να ξέρουμε πάνω κάτω γιατί ψηφίζουμε. Άρθρο 1, παράγραφος 1. Τροπολογία 2 της συγκήτριας. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. Κυρία Λόπε Φοντανιά, πώς ψηφίσατε. 21 ψήφι υπέρ, 19 κατά, 2 αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 13 αποσύρεται. Άρθρο 2, παράγραφος 2. Σημείωση ιότα. Ε, Ι. Τροπολογία 14. Στάινρουκ και Κρίστενσεν. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Από τις πρακτικές μέχρι spacecraft. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές για τα διαστημόπλαια. Ε, δε, υπόλοιπο κείμενο υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 15, μη παραδεκτή. Τροπολογία 16, σε δύο τμήματα. Έκθεση Στάινρουκ. Ε, συγγνώμη, ε, τροπολογία Στάινρουκ, ε, Τανασέσκου, Κρίστενσεν. Πρώτο τμήμα ψηφίζουμε από το Occupation Media Work. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται το υπόλοιπο κείμενο τώρα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Άρθρο 4, παράγραφος 1, σημείο 35, τροπολογία 17 των ιδίων. Πάλι τροπολογία κατά τμήματα. Ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα από το exposed μέχρι το public exposure. Ποιος είναι υπέρ. κατά, αποχές, εγκρίνεται. Το υπόλοιπο κείμενο υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Παράγραφος 3 της ηγετρίας. Ποιος είναι υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 18, μη παραδεκτή. Τροπολογία 4 της ηγετρίας. Ποιος είναι υπέρ. Αφορά το 5 άρθρο. Υπέρ, κατά, αποχές, μάλλον εγκρίνεται αλλά ας το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. 23 ψήφισαν υπέρ και 19 κατά. Εγκρίνεται. Παράγραφος 5. Ποιος είναι υπέρ. Τροπολογία 5. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Άρθρο 6. Παράγραφος 1. Τροπολογία 19. Στάινρουκ και Κρίστενσεν. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η έξι έχει αποσυρθεί ψηφίζουμε για το άρθρο 11 παραγραφος 1 την τροπολογία 20 Στάινρουκ Τανασέσκο Κρίστενσεν ψηφίζουμε σε δύο τμήματα για το πρώτο τμήμα Ποιο είναι υπέρ μέχρι το πρέγνανση κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα το υπόλοιπο κείμενο Ποιο είναι υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. Οι τροπολογίες 21 και 7 έχουν αποσύρθει. Ψηφίζουμε για το άρθρο 12, παράγραφος 2, από παράγραφος 2, σημείο α, την τροπολογία 22 του κυρίου Τσάμπα Όρη. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Επόμενο σημείο, 23, τροπολογία υπέρ, κατά, αποχές, Ηλεκτρονικό έλεγχος για την τροπολογία 23. «43 ψήφισαν, 32 υπέρ, 9 κατά και 2 αποχές». Εγκρίνεται με διαφορά κιόλα. Άρθρο, ε, τροπολογία 24 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 25, Στάινρουκ, Θανασέσκου, Ποιο είναι υπέρ, κατά, αποχέ. εγκρίνεται. Τροπολογία 26 όρη. Ποιο είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 27 το ίδιο υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Για το άρθρο 16, παράγραφος 1, πρότυπο παράγραφος, νέα, Έχουμε προφορική τροπολογία της Γιούτα Στάινρουκ. Ποιος είναι υπέρ? Κατά αποχές. Μάλλον απορρίπτεται, αλλά στο ελέγξουμε καλύτερα. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Ψήφισαν 24 υπέρ και 19 κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 28, Τσάμπα Όρη. Ποιο είναι υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. Τροπολογία 8 τη ηγήτρια. Ποιο είναι υπέρ. Κατά αποχέ απορρίπτεται. 9 τη ηγήτρια υπέρ. Κατά αποχέ απορρίπτεται. 10 τη ηγήτρια υπέρ. Κατά αποχέ απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία Α. 5 ομάδων. Ποιο είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 30, Φιλ Μπένιον, ποιος είναι υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 31, της ηγήτριας, για διαγραφή, ποιος είναι υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 32 της ηγήτριας, υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. Άρθρο 28, παράγραφος 1, τροπολογία 12 της ηγήτριας, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 33, τσαμπαόρι, ποιος είναι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Για το άρθρο 31, παράγραφος 1 ε, συμβαστική τροπολογία β, δύο ομάδων, ποιος είναι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 33, παράγραφος 3, εισαγωγικό τμήμα, τροπολογία 35, Κρίστιν Στάιρο. υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 36 των ιδίων, Ποιο είναι υπέρ, Ηλεκτρονικό έλεγχο θέλετε για το 35. Οκ. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. 20 ψήφισαν υπέρ και 23 κατά. Είχατε απόλυτο δίκιο, απορρίπτεται. Τροπολογία 36 τώρα, των ιδίων. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 37 των ιδίων υπέρ. Κατά Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 38. Τσάμπα όρη. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 39. Το 2 με προφορική τροπολογία. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 40 της συγκήτριας. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 41. Τσάμπα Με προφορική τροπολογία. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 42 του ιδίου. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 43 όροι και πάλι. Με προφορική ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 44 όροι. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 45 του ιδίου. Υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 46 ε, μη παραδεκτή, 47 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 48 φιλμπένιον ποιος είναι υπέρ κατά εγκρίνεται 49 τσάμπα Ποιο ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 50 τσάμπα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 51 μη παραδεκτή 52 προφορική τροπολογία του τσάμπα υπέρ κατά δεν ψηφίσατε. 52. Ποιο είναι υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. Με διαφορά. Τώρα για τις αιτιολογικές σκέψει. Για την αιτιολογική σκέψη 24. Τροπολογία 1. Ποιο είναι υπέρ. Κατά αποχέ. απορρίπτεται. Ψηφίζουμε το σύνολο του κειμένου. Ηλεκτρονικά παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Σαράντα μία ψηφί υπέρ, μία κατά και δύο εποχές. Μία διόρθωση. 40 υπέρ, μία κατά και δύο εποχές γιατί περισσεύει ένας σοσιαλιστής.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 Bien, chers collègues, 22. <coughs> Περνάμε στο σημείο 22 τώρα, αγαπητοί συνάδελφοι. Euh, du rapport de Madame. Έκθεση Όμεν Ρόιτεν. rapport d'initiative sur Έκθεση της Επιτροπής, έκθεση της πρωτοβουλίας. Ατζέντα για επαρκής, ασφαλής και βιώσιμες συντάξεις. Με βάση τον κανονισμό, με βάση τους κανόνες 164 και 161 που προβλέπουν το, τη σειρά ψηφοφορίας και για τις συμβαστικές τροπολογίες που προηγούνται των υπολείπων. Είναι η αυτό που εφαρμόζει και Λομέλεο. Παράγραφο 1. Συμβαστική τροπολογία Α. 5 ομάδων. Ποιο είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 2, τροπολογία 68. Ποιος είναι υπέρ για διαγραφή. Κατά αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος 2 για τη συμβεστική τροπολογία Β. Ποιος είναι υπέρ τριών ομάδων. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 3. Συμβαστική τροπολογία Σ. 5 ομάδων. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 3 Τροπολογία 95 της κυρία Ζουμπέρ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος 4. Συμβεστική τροπολογία δέλτα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συγγνώμη. Παράγραφος Συμβεστική τροπολογία Y ε από τέσσερις ομάδες. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Η 145 έχει αποσυρθεί και ψηφίζουμε την 146 Thomas Handel, που ζητά διαγραφή. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τη συμβαστική τροπολογία ε Ε4 ομάδων υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Μετά την παραγραφό 5, συμβεστική τροπολογία G από 5 ομάδες, Ποιο είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Μετά την παραγράφο 5, τροπολογία 152 τη συγγήτριας και του Ζορς Μπαχ, Ποιο είναι υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονικός έλεγχος παρακαλώ για την τροπολογία 152. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε. Τέλος ψηφοφορίας. 27 ψήφισαν υπέρ, 15 κατά. Εγκρίνεται. 153 τροπολογία των ιδίων. Ποιος είναι υπέρ, κατά αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία F για την παράγραφο 6 από 4 ομάδες. Υπέρ, κατά αποχές. Εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 6 τροπολογία Τζιν Λάμπερτ 161. Τζιν Λάμπερτ και Κορνέλισεν. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 162. Μιναντόρα Κλειβέτη. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 162. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. 20 ψήφισαν υπέρ, 22 κατά. Απορρίπτεται. Παράγραφος 7. Τροπολογία 164. Φρεντερίκ Ταρντέν. Με προφορική τροπολογία. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. 165. Της κυρία Ζουμπέρ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 167. Thomas Τόμας Χέντελ, ποιος είναι υπέρ. Χέντελ, sorry, όχι μαν. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Να ψηφίσουμε την 171 της κυρίας Γιαζοβίατσικα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 7, τροπολογία 172, Μπέκερ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 173 του κυρίου Τρεμόσα Υπαλσέλς. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 174 της κυρία Ζουμπέρ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος 8. Σάντσες. Βιζότο Ποιος είναι υπέρ. Ζητά διαγραφή κύριε Βιζότο. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία H. 5 ομάδων υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 8 έχουμε την τροπολογία 100 87 του κυρίου Μπέκερ με προφορική τροπολογία των σοσιαλιστών. Ποιος είναι υπέρ της 187 όπως έχει τροποποιηθεί. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 187. Tout le monde a pu voter. Le vote est clos. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. 27 υπέρ 12 κατά, 3 αποχές, εγκρίνεται σαφέστατα. Παράγραφος 9. Συμβαστική τροπολογία HH με 4 ομάδων υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά την παραγραφό 9, τροπολογία 199. Μπέκερ. Ποιος είναι υπέρ. 199 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Θέλετε ηλεκτρονικό έλεγχο για την 199 του κυρίου Μπέκερ. Αυτή την αίσθηση έχω. Ωραία. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 199 του κυρίου Μπέκερ. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι ωραία. 6 υπέρ, 32 κατά, 3 αποχές. Μάλλον 33 ψηφί κατά. Hey, Κυρία Χάρκιν, εσεί τι ψηφίσατε. Α, 7 υπέρ τότε, 32 κατά, 3 αποχές. Απορρίπτεται ούτως ή άλλως. Μετά την παράγραφο 9, τροπολογία 200 του Τόμας Χέντελ, Ποιο είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Μετά την παράγραφο 9, τροπολογία 202 του ιδίου υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος 10, τροπολογία συμβαστική γιώτα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 10, τροπολογία 210 του Σέρτζο Κοφεράτη. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές Ηλεκτρονικός έλεγχος για τη 210. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. 19 ψήφισαν υπέρ και 22 κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 11. Δύο τροπολογίες για διαγραφή. 212 Νταρντέν και 213 της κυρίας Μπιτζότο. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. Ψηφίζουμε την τροπολογία 2.14 του Thomas Handel. Ποιος είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 215 Ζουμπέρ, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Μετά την παράγραφο 11, τροπολογία 218. τώρα κλειβέτη με προφορική τροπολογία. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, Απορρίπτεται. Συμβαστική 12, ε, J, παραγραφό 12, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Μετά την παραγραφό 12, τροπολογία 226 του Τόμας Χέντελ, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Μετά την παραγραφό 12, τροπολογία 227, καταπίπτει. Και περνάμε στη βεστική τροπολογία K, 5 ομάδων. Ποιο είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 13, τροπολογία 232 του κυρίου Μπέκερ. Ποιο είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 233, Τόμας Χέντελ. Ποιο είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 2.36 Μπέκερ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.37 Χέντερ υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για τη 2.37 άρχεται ψηφοφορία Ψήφισατε όλοι. 21 ψηφί υπέρ, 22 κατά απορρίπτεται. Δύο 14 ε, διαγραφή υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Δύο 14 είπα λέει πρόεδρος. Αχ, δυσλεξία με έχει πιάσει. Συμβαστική τροπολογία μη. Ποιο είναι υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται η συμβαστική τροπολογία μη. Μετά την παράγραφο 14, τροπολογία μη από πέντε ομάδες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 15. Τροπολογία 258 του Τόμας Χέντελ. Ζητά διαγραφή. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβεστική τροπολογία ο μικρόν υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Για την παράγραφο 16. Τροπολογία 263 του Φρεντερικ Νταρντέν. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Οι 264 και 265 αποσύρονται. 266 Kinga Gunts Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Για την παραγράφο 17, συμβαστική τροπολογία P από 5 ομάδες, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 17, συμβαστική τροπολογία L από 5 ομάδες, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ε, 281 Νταρντέν, η συγκεντρία είναι κατά. Ποιος είναι υπέρ της 281. Κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για την 281. Παρακαλώ, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. 26 υπέρ 17 κατά εγκρίνεται. 283 της κυρίας Μακιντάιρ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Για την παράγραφο 19 συμβεστική τροπολογία Q. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος R. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία συμβαστική τροπολογία S ποιος είναι υπέρ στην παράγραφο 21 κατά αποχές εγκρίνεται για την παράγραφο 22 τροπολογία 30, 300 συγγνώμη για Ζωβιέτσικα ζητά διαγραφή υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ψηφίζουμε την 301 της κυρίας Ζουμπέρ υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Μετά την 22, τροπολογία 302 της συγκέντριας και του Ζορς Μπάχ υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Μετά την 22, τροπολογία 303 του Ζαμπιέρ Οντί, με προφορική τροπολογία, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Σε συμβαστική τροπολογία τι, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Για την αιτιολογική σκέψη α, στο έκτο εδάφιο, τροπολογία 12 καταπίπτει. Αιτιολογική σκέψη Β, συμβαστική τροπολογία ΤΑΦ, 5 ομάδων υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά την αιτιολογική σκέψη Β, τροπολογία 24 της κυρίας Μακιντάιρ με προφορική τροπολογία της ιδίας. Ποιο είναι υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία U για την αιτιολογική σκέψη C. Ποιος είναι υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. Μετά την αιτιολογική σκέψη C, τροπολογία 29 της κυρίας Γεζοβιέτσκα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Μετά την αιτιολογική σκέψη C, τροπολογία 30 του Τόμας Χέντελ. Σε τρία τμήματα ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα. από τους δημογραφικούς δείκτες μέχρι κοινώς αποδεκτό. Ποιος είναι υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα καταπίπτει, αν δεν κάνω λάθος, και το ίδιο ισχύει για το τρίτο τμήμα. Γιατί ψήν που υπάρχει δεαρφορός εκ τούτου συνδυάζεται με το προηγούμενο τμήμα. Αιτιολογική σκέψη Δ. Συμβαστική τροπολογία Β από πέντε ομάδες. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 35 το Τόμας Χέντελ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία ε. ε συμβαστική τροπολογία μάλλον W για το διαλογική σκέψη ε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 41. Τόμας Χέντελ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος γιατί δεν έχουν ψηφίσει όλοι. Τροπολογία 41, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. 20 υπέρ, 21 ψήφι κατά, χωρίς αποχές. Οπότε καταπίπτει η τροπολογία 41. Μετά την αιτιολογική σκέψη ε, τροπολογία 44 του Τόμας Χέντελ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ε, αιτιολογική σκέψη F, συμβαστική X, ε, X, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Μετά την αιτιολογική σκέψη F, Πάμε στην τροπολογία 53 της συγγήτριας και του Ζορς Μπαχ. Ψηφοφορία κατά τμήματα. Ψηφίζουμε το κείμενο χωρίς το at a fast pace, με γοργό ρυθμό. Ποιος είναι υπέρ του πρώτου τμήματος, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και ποιος θέλει να πάει με γοργό ρυθμό, υπέρ, το δεύτερο τμήμα δηλαδή, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Μετά την αιτιολογική σκέψη F, τροπολογία 55 του κυρίου Πουπάκη. Ποιο είναι υπέρ, κατά, απόχέ εγκρίνεται. Μετά την αιτιολογική σκέψη F, τροπολογία 56 της συγκίτριας και του Ζόρς Μπαχ. Ποιο είναι υπέρ, κατά, Αποχέ εγκρίνεται. Μετά την F πάλι 57 τροπολογία του Φιλίπ Νταρντέν υπέρ κατά απόχέ. απορρίπτεται για το θεωρώντας. Μετά το θεωρώντας 7, τροπολογία 1 του ιδίου, υπέρ. Α, δεν είχα ενημερωθεί για την απόσυρση. Οπότε μετά το θεωρώντας 8 ψηφίσουμε τροπολογία 2 του Τόμας Χέντελ. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, κατά, αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 2 άρχιτη ψηφοφορία ψηφίσατε όλοι τέλος ψηφοφορίας 22 υπέρ 19 κατά εγκρίνεται μετά το θεωρώντας 8 τροπολογία 3 του Φρεντερικ Νταρντέν ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Περνάμε τώρα στις γνωμοδοτήσεις των επιτροπών. Τροπολογίες 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 κτλ. κτλ, μέχρι την 70 της Οικονομικής Επιτροπής εμπίπτουν στην αποκλειστική μας αρμοδιότητα, γι' αυτό και δεν θα τις ψηφίσουμε. Αφορούν το δεύτερο πυλώνα. Αντίθετα θα πρέπει να ψηφίσουμε κάποιους παραγράφους για τους οποίους ισχύει κοινή αρμοδιότητα. Και μετά την ψηφοφορία αυτές οι παράγραφοι θα ενσωματωθούν σε κάποια τμήματα της έκθεσης. Αυτό θα το φροντίσει η συγγήτρια με τους πιο δισηγητές για το ποιο είναι το κατάλληλο σημείο να ενσωματωθούν οι, οι παράγραφοι αυτές. Παράγραφος 4. Ποιος είναι υπέρ της εικόν, εκών. Υπέρ της 4. Η εισηγήτρια είναι κατά πάντως. Ποιος είναι υπέρ. Ποιος είναι υπέρ, λέω, της παραγράφου 4 της Οικονομικής Επιτροπής. Κατά τώρα. Αποχές. Απορρίπτεται η παράγραφος 4. Παράγραφος 10 της Οικονομικής Επιτροπής. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την παράγραφο 10 της ΕΚΟΝ. Οι σοσιαλιστέ στην ΕΚΟΝ είναι κατά του ΕΛΚ. Τέλος ψηφοφορίας. 21 ψήφισαν υπέρ. Κυρία, Κυρία Χάρκιν, τι ψηφίζετε εσεί. Μαριάν. Ωραία. 22 υπέρ 17 κατά. Μηδέν αποχές. Η παράγραφος 10 ε, εγκρίνεται. 11 τώρα, Επιτροπή Έκων. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 22 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ένα τμήμα της παραγράφη 25 από έκον υπέρ κατά υπέρ ξανά, κατά αποχές ξεκάθαρα εγκρίνεται 37 ολόκληρη υπέρ κατά αποχές επαλήθευση για την παράγραφο 37 της ΕΚΟΝ. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. 25 υπέρ 16 κατά εγκρίνεται. Παράγραφο 47. Έκον πάλι υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. Ένα τμήμα της παραγράφου 49 της Επιτροπής ΕΚΟΝ. Επαλήθευση για τη 47. Έναρξη ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. 25 υπέρ 16 κατά δίκιο είχατε. Εγκρίνεται η παράγραφος 47. Τώρα, ένα τμήμα της 49 υπέρ. Κατά αποχές θα ελέγξουμε την παράγραφο 49. Ηλεκτρονικός έλεγχος παρακαλώ. Πέρας. 25 υπέρ 16 κατά. Επίσης εγκρίνεται. Κυρία Μενρόιτερ. Κοιτάξτε, θα ήθελα να πω στους ε, συναδέλφους μου ότι εγώ δεν είμαι κατά του περιεχομένου, αλλά οι τροπολογίες της Επιτροπής ΕΚΟΝ ήδη περιλαμβάνονται στις εκθέσεις. Αυτός λοιπόν είναι ο λόγος που διαφωνούμε, ότι είναι λάθος, μεγάλο λάθος, το γεγονός ότι καλούμεθα να ψηφίσουμε για αυτές τις ε, παραγράφους. Θέλω λοιπόν να πω στους ε, συναδέλφους μου ότι εφόσον υπάρχουν νέα στοιχεία ε, πρέπει να τα εγκρίνουμε και συμφωνώ από αυτό. Αλλά αυτό που κάνουμε τώρα είναι ε, τρελό. Το ίδιο ισχύει και για την ε, Επιτροπή Μεταφορών. Ε, των γυναικών, με συγχωρείτε. Συγγνώμη, έχουμε την άποψη της εισηγήτριας, ε, όμως κάναμε ένα προσεκτικό έλεγχο και ως ήθιστε Έλεγξαμε ποιε ήταν οι παραγραφοί που καλύπτονταν και ποιε όχι. Στην έκθεση το Μασμάν τη Επιτροπής ΕΚΟΝ κρίναμε ότι μία σειρά τροπολογιών όντως καλύπτονταν και ω εκ τούτου δεν ε, αναγράφονται στον κατάλογο ψηφοφορίας. Παραγραφή 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 47, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 62, 72, 74 και 75. Ε, σας τα λέω όλα αυτά για να σας εξηγήσω ότι εκτεταμένα ασχοληθήκαμε με το ζήτημα. Αλλά έχουμε μία δεκαπενταριά παραγράφους που βλέπουμε ότι δεν έχουν καλυφθεί. Και για, εσείς έχετε για το σύνολο αυτών των παραγράφων εκδώσει, ε, συγγνώμη, υποδείξει αρνητικό πρόσημο για, τις, ε, για την ψηφοφορία. Ε, θα συνεχίσουμε από εκεί που σταματήσα. Όπι, κυρία Μπάστος, θα ήθελα να μάθω κάτι, διότι λάβαμε με μεγάλη καθυστέρηση τον κατάλογο ψηφοφορία. Είναι ο ίδιο που ισχύει για την ψηφοφορία στην Επιτροπή Γυναικών. Απάντηση. Μην ανησυχείτε. Τα ίδια ισχύουν και για την Επιτροπή Γυναικών. Έχουμε μία εικοσαριά παραγράφους από την Επιτροπή Γυναικών που μπορούμε να ψηφίσουμε διότι δεν καλύπτονται από την γνωμοδότηση της κυρίας Όμενε Ρόιτεν ούτε και από τις τροπολογίες που μόλις ψηφίσαμε. Ιδού. Εντάξει. Είστε όλοι ικανοποιημένοι τώρα. Τι ποιο πρόβλημα υπάρχει ακόμα. Voilà. Moi, écoutez, euh, Λοιπόν, εγώ ήλεγξα το θέμα με την ε, γραμματεία. Ποιε είναι οι θέσει των μεν και των δε και καταλήξαμε στο ότι είναι απολύτω ορθός ο κατάλογος ψηφοφορία που έχετε ενώπιον σα. Αν κάποιε πολιτικέ ομάδε κρίνουν ότι πρέπει να επιφέρουμε ε, τροποποιήσει στον κατάλογο, α επομιστεί η πολιτική ομάδα που έχει αμφιβολίε την ευθύνη και σε επανέλθουν στην Ολομέλεια. Εμεί θα συνεχίσουμε την ψηφοφορία μα σε κάθε περίπτωση. Ήμασταν στην παράγραφο 57, Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών. Υπέρ και σας υπενθυμίζω ότι είναι κατά η συγγήτρια. Η συγγήτρια όμως της Επιτροπής ΕΚΟΝ θα ήθελε πολύ να την ψηφίσουμε αυτή την τροπολογία. Ποιοι είναι υπέρ της 57. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ε, χάρη και η συγγήτριά μας, θα την αχαρεί η συγγήτρια της ΕΚΟΝ. 58 τώρα, υπέρ. Κάτα. Άποχες. Απορρίπτεται. 59. Πάλι της ΕΚΟΝ, υπέρ κατά αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται. Αντιπρόεδρε, για σας το έκανα. 71 της έκον υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, απορρίπτεται. Καλά, καλά, καλά, καλά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Έρχεται για την 71 και η κυρία Χάρκιν ε, ψηφίζει υπέρ. Πέρας. 27 προς 15, ξεκάθαρα εγκρίθηκε. 73 της έκον υπέρ. Κάτα. Άποχες. Εγκρίνεται. Ήμκο. Εδώ έχουμε να ψηφίσουμε μόνο την τροπολογία 5, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην Επιτροπή Γυναικών. Εδώ τι έχουμε να ψηφίσουμε. Euh, je, je est-ce que quelqu'un voit un inconvénient est-ce que nous suivons la liste de vote Υπάρχουν ενστάσεις, μπορούμε να ακολουθήσουμε τον κατάλογο ε, ελαφρώ αντίστροφα, δηλαδή να ψηφίσουμε πρώτα τις αιτιολογικές σκέψεις και μετά τις παραγράφους. Ωραία. Ε, αποκλίνουμε από τους κανόνες μας. Ε, το ΣΕ της Επιτροπής Γυναικών υπέρ. Κατά. Άποχες. Έλεγχο. Για το εκτιμώντα ε, την αιτιολογική σκέψη C. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 24 προς 17 και μία αποχή. Εγκρίνεται. Το D τώρα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Το K. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. L. Υπέρ. Κατά. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Έλεγχος. Άρχεται. Πέρας. 25 προς 17. Εγκρίνεται. M υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Εκτιμώντας N υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. O υπέρ. Κατά αποχές, απορρίπτεται. Παράγραφος 2, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 52 το πρώτο τμήμα μέχρι το μένεις Applied, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, το υπόλοιπο, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η 7, παράγραφος 7, φαμ, σε δύο τμήματα. Το πρώτο μέχρι το labor market υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται το υπόλοιπο υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Έλεγχος για το δεύτερο τμήμα της παραγράφου 7 άρχεται. Πέρας. 25 ψήφοι υπέρ προς 17 κατά, μία αποχή, εγκρίνεται επίσης. Η παράγραφος 8, φαμ, υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. 12, Επιτροπής Γυναικών υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. 17, της ίδιας Επιτροπής υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτεται. 20 της ίδιας Επιτροπής, έλεγχος για τη 17 παρακαλώ. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. 25 προς 17 εγκρίνεται. 20 της ίδιας Επιτροπής υπέρ. Κάτα έλεγχος για την 20. Ψήφισαν όλοι. πέρας. 25 προς 17 επίσης εγκρίνεται. 23 της ίδιας Επιτροπής υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 30 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 31 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Το σύνολο τώρα με ηλεκτρονική ψηφοφορία για την έκθεση. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας. 32 ψήφοι υπέρ, 4 κατά 6 αποχές. Συγχαρητήρια στην εισηγήτριά μας. Μην ναι, πάνω, πάνω. Μη φύγετε. Μη, μη, μη, μη, καθίστε εδώ. Nous avons encore un vote. Έχουμε άλλη μια ψηφοφορία. Σημείο 23. Και όμως Ρόιτεν, τι θέλετε. Μα μη φύγετε, έχουμε άλλη μία ψηφοφορία και χρειαζόμαστε ειδική πλειοψηφία. Καθίστε στις θέσεις σας παρακαλώ. Κυρία Όμεν δύο παρατηρήσεις έχω. Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνεργάστηκαν ε, γιατί, μαζί μας γιατί είναι καλό το αποτέλεσμα. Ευχαριστώ λοιπόν όλους του συναδέλφους. Δεύτερον, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί γιατί στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων είναι καλό το αποτέλεσμα, το περιεχόμενο δηλαδή, αλλά αυτά που ψηφίσαμε για την Επιτροπή Έκων και ε, Γυναικών ως επιτοπλίστων ή καλύπτονται από την έκθεση ή αντίκειται στην έκθεση. Οπότε ε, η Γραμματεία παρακαλείται να δει με ποιο τρόπο θα προχωρήσουμε πριν πάει στην Ολομέλεια. Εντάξει, το είπαμε, κυρία Ομένερο, ήταν είπαμε ότι είναι ευθύνη των πολιτικών ομάδων. Και εμεί τα ψηφίσαμε γιατί δεν καλύπτονταν αυτά τα σημεία που μόλι ψηφίσαμε. Σημείο 23. Α ακούσουμε την κυρία Χάρκιν. Ε, πρόκειται για τη διαπραγματευτική εντολή για το Ταμείο Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση 2014-2020 και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 7η και 8η Φεβρουαρίου. κύρωσε την ε, απόφαση για το ταμείο αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, πολύ σύντομα να πω για να ξέρετε κι εσείς ότι η απόφαση που ελήφθη είναι να συνεχιστεί αυτό το Ταμείο της Παγκοσμιοποίησης ε, ε, με περιορισμένο βέβαια προεπολογισμό των 150 εκατομμυρίων το χρόνο. Ε, υπάρχει κάποια ανασφάλεια σχετικά με το μέλλον του Ταμείου στις 22 Μαρτίου. Η Αρμόδια Επιτροπή ελπίζουμε ότι θα οριστικοποιήσει τις απόψεις της σχετικά με τα επίμαχα θέματα του Ταμείου και στις 27 Μαρτίου ε, το, η Κορεπέρ θα ασχοληθεί και αυτή με το θέμα με στόχο να εκδώσει εντολή έτσι ώστε να υπάρξουν διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Θέλω λοιπόν απλά να πω ότι εμείς πρέπει να ψηφίσουμε για να δώσουμε ένα ε, θετικό μήνυμα προς το Συμβούλιο. Πρέπει οι διαπραγματεύσεις να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το Σεπτέμβριο αν θέλουμε το Ταμείο αυτό να αρχίσει να λειτουργεί ε, την 1η Ιανουαρίου. Αυτός λοιπόν είναι ο στόχος της ε, ψηφοφορίας που λαμβάνει η χώρα σήμερα. Ωραία, σας ευχαριστούμε. Θα ψηφίσουμε με ηλεκτρονική ψηφοφορία την ε, αίτηση διαπραγματευτικής ε, εντολής ε, για την έκθεση που ψηφίσαμε στις 6 Νοεμβρίου και της κυρίας Χάρκιν. Παρακαλώ, ψηφίστε. Ψήφισαν όλοι. Περάς. 37 ψήφοι υπέρ, μία κατά και μία αποχή. Η διαπραγματευτική ομάδα θα απαρτίζεται από μένα με την ιδιότητα της Προέδρου, την κυρία Χάρκιν με την ιδιότητα της εισηγήτριας, σκιώδης του Έλκιν η κυρία Μπάουρ, Νταρντάν σκιώδης ε, των Σοσιαλιστών, η κυρία ένα από τους Πρασίνους, ε, Τσούμπερ Γκούε, ε, Γκάπ Μόρα από τους Συντηρητικούς και Πιτσότο από την Ευρώπη της Ελευθερίας και της Δημοκρατίας. Και ολοκληρώνουμε έτσι και αυτό το σημείο της ε, ε ημερήσιας διάταξης και φτάνουμε στο σημείο 24 ε, για την εξέταση 517 τροπολογιών που κατατέθηκαν για την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πρόταση κανονισμού σχετικά με το Ταμείο Ενίσχυσης των Απόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης η συγγήτριά μας, Έμερ Κοστέλο, θα πάρει τον λόγο. Σας ακούμε. Thank you very uh, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και όπως ε, πολύ σωστά είπατε είχαμε 570 ε, περίπου τροπολογίες στην ε, πρόταση που κατατέθηκε στην Επιτροπή. Νομίζω λοιπόν ο μεγάλος αριθμός των ε, τροπολογιών που κατατέθηκε καταδεικνύει το ενδιαφέρον που υπάρχει για το πρόγραμμα αυτό και τη δέσμευση των ανθρώπων απέναντι στο πρόγραμμα. Ε, το πώς οι άνθρωποι δεσμεύονται να βελτιώσουν την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τροπολογίες μας διατέθηκαν μόλις τη Δευτέρα. Ε, πρέπει να σας πω ότι εγώ δεν μπόρεσα να μπω σε λεπτομέρειες. Ε, προσβλέπω στο να τις ε, επανεξετάσω λεπτομερώς από κοινού με τους ε, σκιώδεις. Με την πρώτη εξέταση των τροπολογιών εντόπισα ότι υπάρχει ένα ευρύ κοινό πεδίο και θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμβαστικές προτάσεις αρκετούς τομείς που σημαίνει ότι οι τομείς αυτοί είναι οι εξής παραδείγματο χάρη να γίνεται καλύτερη αναφορά στο χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Επίσης, ε, ε, να γίνεται καλύτερη αναφορά στου ε, κοινωνικά αποκλεισμένου, να υπογραμμιστεί η σημασία του να προσφέρονται ποιοτικά τρόφιμα και μάλιστα υγιή τρόφιμα να συμπεριληφθούν τα σχετικά κατόφλια φτώχεια, να στηριχθούν προγράμματα, εθνικά προγράμματα επισητιστικής βοήθειας και επίσης να υπάρξει συνεργασία με τους μη κυβερνητικές οργανώσεις ε, ε, έτσι ώστε ε, να προαχθεί στην εργασία αυτή, να αρθούν ε, τα εμπόδια που εμποδίζουν ε, την διανομή τροφίμων από τις αλυσίδες τροφίμων. Επίσης, να εξευρεθούν ορισμοί, αυτό είναι πολύ σημαντικό και είναι σημαντικό να υπάρξουν και κάποιες τροπολογίες που αφορούν στην διευκρίνηση των ολογιών σχετικά με τους τελικές αποδέκτες όλων αυτών των ευνοϊκών διατάξεων. Αυτό που ενδιαφέρει επίσης είναι να προάγεται η ανθρώπινη αξιοπρέπεια και να αποφεύγεται ο στιγματισμός όλων των αποδεκτών της ε, βοήθειας σε τρόφιμα. Είναι σημαντικό ε, να περιοριστεί η σπατάλη των τροφίμων. Αυτό διατρέχει ως κοινό στοιχείο όλες τις ε, τροπολογίες. Εξάλλου πολλά μέλη αναφέρουν ότι είναι απαραίτητο η ύπαρξη του Ταμείου να μην ε, επικαλύπτει, να μην συγκαλύπτει την ανάγκη να υπάρχουν και άλλα εθνικά προγράμματα. Πολλές λοιπόν ε, τροπολογίες ε, αναφέρουν ότι είναι απαραίτητο να υπάρξουν διαδικασίες απλούστευσης και μάλιστα και απλουστευμένες διαδικασίες εξέταση των θεμάτων. Υπάρχουν κάποια ψηφίσματα που αναφέρονται σε πρώην ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, παραδείγματος χάρη για τους αστέγους. Επίσης υπάρχει μία σωρά, <clears throat> σειρά τροπολογιών που αναφέρονται στα συνοδευτικά μέτρα και μία σειρά τροπολογιών επιθυμεί να διευκρινίσει ε, το τι ακριβώς είναι οι πολίτες ε, που ε, στερούνται σχεδόν τα πάντα από πώς ορίζονται αυτοί σε αντίθεση και σε διαχωρισμό από τους υπόλοιπους. Κατόπιν, το θέμα των αλυσίδων παροχής ε, τροφίμων. Εδώ πάλι το θέμα των ποιοτικών τροφίμων, των υγιών ε, τροφίμων και ε, την χρήση των ντόπιων προϊόντων. Μία σειρά τροπολογιών εξετάζει <clears throat> τους τομείς όπου μπορούμε να επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και πώς αυτά μπορούν να στηριχτούν από μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα που έχει σχέση με την ανταλλαγή πληροφοριών. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες ενδιαφέρουσες απόψεις οι οποίες εκφράζονται μέσω αυτών των τροπολογιών. Ορισμένες από τις τροπολογίες επίσης εξετάζουν το αίτημα της Επιτροπής να ε, εξετάζονται οι συνεργασίες ε, κυρίως όσον αφορά συνεργασία ε, με κοινωνίες ε, των πολιτών. Ε, μία σειρά τροπολογιών. Επίσης, ζητά από την Κομισιόν να αναφέρεται τακτικά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο και νομίζω ότι είναι σημαντικό το Κοινοβούλιο να διδραματίσει σημαντικό ρόλο στον έλεγχο του προγράμματος. Ορισμένες από τις τροπολογίες επίσης εξετάζουν ε, το ότι πρέπει να διασφαλιστεί, το ότι οι αρχές κομισιών ε, πρέπει να αναφέρουν την πρόοδο, ε, να προβαίνουν και σε βελτιώσεις εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο. Εξάλλου, στεναρή υποστήριξη προσφέρεται σε τομείς που έχουν σχέση με συνοδευτικά μέτρα όπου διασφαλίζεται ότι δεν θα πρέπει όλες οι συνεργασίες ε, να προβαίνουν ε, και να λαμβάνουν ε, συνοδευτικά μέτρα. Αυτό αφορά βέβαια τις ΜΚΟ και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Τώρα, όσον αφορά στις διατάξεις εξαίρεσης και τις διατάξεις αξιολόγησης, Νομίζω ότι κατατέθηκαν και κάποιες τροπολογίες και σχετικά με αυτό. Υπάρχουν ε, εξάλλου αρκετοί ε, τομείς ε, όπου προκύπτει διαφωνία ανάμεσα στα μέλη και αυτά πρέπει να συζητηθούν περαιτέρω σε συναντήσεις των σκιωδών εισηγητών. Πρώτον, όσον αφορά όλο αυτό το θέμα της συγχρηματοδότησης. Υπάρχουν αρκετές τροπολογίες που ζητούν χρηματοδότηση 100% από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ άλλες πάλι στηρίζουν την πρόταση Κομισιόν για τη συγχρηματοδότηση. Υπάρχουν και άλλες προτάσεις ε, που έχουν σχέση με τη συγχρηματοδότηση και ζητούν είτε ε, προοριτική συγχρηματοδότηση είτε κάτω από ορισμένε συνθήκες. Ε, πρέπει να εξεταστούν ε, ιδιαίτερα αυτά τα θέματα. Κατόπιν υπάρχει και μία σειρά τροπολογιών που καλεί ε, τα κράτη-μέλη και ε, όπου προβλέπεται ότι η συμμετοχή των κρατών μελών ε, θα είναι προαιρετική. Άρα δηλαδή και αυτό πρέπει να το συζητήσουμε λεπτομερώς. Ανέφερα ότι στην συνάντηση που παρουσιάστηκε για έκθεση την περασμένη Δευτέρα ετέθη το θέμα της προαιρετικής συμμετοχής και είπαμε είναι σημαντικό να διασφαλίζεται ότι το Ταμείο ε, θα οχυρώνεται, θα οχυρωθεί για το πρόγραμμα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό εφόσον επιθυμούμε να υπάρχει προαιρετική συμμετοχή και εφόσον εγκριθεί η συμμετοχή αυτή να διασφαλίσουμε ότι η χρηματοδότηση για τις ε, συμμετέχουσες χώρες. Τρίτον, υπάρχουν ε, κάποιες ε, τροπολογίες που καλούν το Ταμείο να στηρίζει μόνο εθνικά προγράμματα τροφίμων. Και αυτό λοιπόν συζητήθηκε λεπτομερώς στην δημόσια κρόση που είχαμε στις 23 Ιανουαρίου και υπήρξε στεναρή υποστήριξη από πολλές οργανώσεις ε, κοινωνίας των πολιτών. Στηρίζουν αυτές ε, τους ευρύτερους στόχους του προγράμματος και ε, θεωρούν ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει η η απαραίτητη ευελιξία στο εφαρμοζόμενο πρόγραμμα. Κατόπιν υπάρχει μια τροπολογία που λέει ότι ε, θα πρέπει να επιβληθούν ε, κάποιες, ε, να εισαχθούν κάποιες διατάξεις σχετικά με την, τα τρόφιμα που περισσεύουν και που πετιούνται. Υπάρχουν κάποιες τροπολογίες σχετικά με τον προϋπολογισμό του προγράμματος. Μερικές εξ αυτών μιλούν για 3,5 δις, μια άλλη τροπολογία αναφέρεται σε 5 δις. Εγώ θεωρώ ότι ε, πολλοί δεν ικανοποιήθηκαν στην Επιτροπή μας με όλα αυτά. Τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο υπήρχαν κάποιες διαφωνίες για τον προπολογισμό και τα πραγματικά στοιχεία του προπολογισμού έχουν άμεση σχέση με το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και φεύγουν εκτός των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής μας, δυστυχώς. Καταλαβαίνω όμως τις ανησυχίες ε, των μελών που επιθυμούν να έχουν αυξημένα κονδύλια. Ένα άλλο θέμα έχει σχέση ή είναι εκείνο που θα προκαλέσει συζητήσεις με τους ε, σκιώδεις, δηλαδή οι τροπολογίες που αναζητούν μια σειρά διαφορετικών ε, δικτών. Ε, υπάρχει μια σειρά προτάσεων για τους δίκτες που πρέπει να χρησιμοποιούνται όπως παραδείγματο χάνει το ποσοστό του πληθυσμού που είναι κάτω από την γραμμή της φτώχειας. Άλλοι δείκτες είναι οι δείκτες που έχουν σχέση με τη φτώχεια ε, που έχουν σχέση με το ποσοστό ανθρώπων που κινδυνεύουν ε, να διολυστήσουν σε επίπεδο φτώχεια. Υπάρχει λοιπόν μια ολόκληρη σειρά θεμάτων που ε, έχουν σχέση με δείκτες. Ένα άλλο θέμα το οποίο εμφανίστηκε στις τροπολογίες έχει σχέση με τα μεταβατικά μέτρα. Τα μέλη ανησυχούν, εξέφρασαν την ανησυχία τους για το ότι το πρόγραμμα δεν θα μπορέσει να εφαρμοστεί μέχρι την 1η Ιανουαρίου του 2014. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό οι οργανώσεις που αυτή τη στιγμή συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα ε, δεν θα πρέπει να κινδυνεύσουν να χάσουν τα κονδύλια τους. Ε, γι' αυτό λοιπόν υπάρχει μια σειρά προτάσεων που εξετάζουν ε, και αυτό το θέμα. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει και εμείς να το εξετάσουμε ε, διεξοδικά. Υπάρχει μία τροπολογία που κατά την άποψή μου ε, λέει ότι η πρόταση πρέπει να απορριφθεί. Εγώ την απορρίπτω αυτή την πρόταση γιατί πιστεύω ότι τα στοιχεία που προέκυψαν από την ακρόαση και από τις διαβουλεύσεις μας με τους ε, φορείς της κοινωνίας των πολιτών και τα, οι απόψεις που εξέφρασαν τα περισσότερα μέλη στις τροπολογίες ή μέσω των τροπολογιών που κατέθεσαν καταδεικνύουν ότι είναι απαραίτητο η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιδείξει αλληλεγγύη με τους ε, στερημένους, ε, με αυτούς ε, που πραγματικά έχουν ανάγκη, που χρειάζονται τα, τις τράπεζες αυτές των τροφίμων, αυτά τα παντοπολία τροφίμων, γιατί οπωσδήποτε πρέπει να συνεχιστεί το πρόγραμμα. Αυτά λοιπόν εν ολίγης πάρα πολύ γρήγορα σχετικά με τις τροπολογίες που λάβαμε και όπως σας είπα υπάρχει ένα τεράστιο περιθώριο ε, επίτευξης συμφωνίας. Έχουμε κανονίσει μια συνάντηση των συντονιστών για την επόμενη εβδομάδα και θα συζητήσουμε τις ε, τροπολογίες τον Απρίλιο. Ελπίζω λοιπόν να οργανωθούν και άλλες ε, συναντήσεις ε, με τους σκιώδεις συγητές μέχρι την επόμενη συνάντησή μας. Ευχαριστώ όλους για τη βοήθειά τους. Νομίζω ότι οι τροπολογίες που έχουμε μας προσφέρουν τη βάση για να προετοιμάσουμε ένα καλό σταθερό πρόγραμμα και πιστεύω ότι τελικά αυτό που θα παρουσιάσουμε ε, θα εξυπηρετήσει, θα υπηρετήσει τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα διαπιστώσατε ότι το Συμβούλιο συζητάει το πρόγραμμα παράλληλα με το Κοινοβούλιο. Τα 2,5 δις ε, συμφωνήθηκαν ε, για το Φεβρουάριο Γνωρίζουμε βέβαια ότι ακόμα υπολείπονται πολλές συζητήσεις και διαπραγματεύσεις σε επίπεδο Συμβουλίου. Εμείς λοιπόν ε, θα παρακολουθήσουμε την εξέλιξη των προγραμμάτων εκ του σύναγης. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε. Ο Τσαμπαόρη είναι ο πρώτος που θα πάρει το λόγο και στη συνέχεια η Μαρία Χάρκιν. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, Επιτρέψτε μου να εκφράσω την ευγνωμοσύνη και τις ευχαριστίες μου προς την κυρία Κωστέλιο. Είμαι σίγουρος ότι ήταν δυσχερές το έργο της. Αυτό που ενδεχομένως θα μπορούσε να το διευκολύνει σχετίζεται με τους βασικούς άξονες που μας βρίσκουν σύμφωνους ναι μεν, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις παράλληλες συζητήσεις που γίνονται στο Συμβούλιο για το Ταμείο Απόρων. Διότι αμφισβητείται ακόμη και η μελλοντική ύπαρξη του Ταμείου από κάποιους. Αυτό που ελπίζουμε είναι να λάβουμε μια επιβεβαίωση από το Συμβούλιο ότι προτίθεται να εξακολουθήσει να εξασφαλίζει τη χρηματοδότηση του Ταμείου. Θα ήθελα να εκφράσω την υποστήριξή μου για την πλειοψηφία των επιμέρους σημείων της έκθεσης. Βεβαίως θα υποβάλω κάποιες τροπολογίες ε, με στόχο να αυξηθεί το ύψος της βοήθειας προς τους πλέον απόρους και να ε, μειωθεί κατά τι η χρηματοδότηση των καπαόμικρων. Μας ικανοποιεί το ποσοστό της βοήθειας, όπως το προτείνει η εισηγήτρια. Δεν μπορούμε ε, χωρίς κανένα αντίκρισμα να ε, παρέχουμε αυτή τη βοήθεια. Ο στόχος μεταξύ άλλων είναι να ευαισθητοποιηθούν τα κράτη-μέλη σε σχέση με τις ανάγκες των απόρων. Τα κράτη-μέλη λοιπόν θα πρέπει να συνδράμουν μέσω του Ταμείου αυτού. Ως προς τον εθελούσιο χαρακτήρα της δράσης αυτού του Ταμείου, βλέπουμε μια διαχωριστική γραμμή ε, που χωρίζει τις κυβερνήσεις σε δύο στρατόπεδα. Θα καταστεί υποχρεωτική η βάση ή θα παραμείνει εθελοντική για την λειτουργία του Ταμείου. Περιπλέκεται δε η κατάσταση διότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο θα χρηματοδοτήσει ένα κομμάτι αυτού του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τους οπόρους προς το παρόν. Ένα τμήμα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, επιθυμεί σε εθελούσια βάση να παρέχεται η βοήθεια. Άρα αυτό το ζήτημα δεν έχει κλείσει και θα πρέπει να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυ τις διαπραγματεύσεις που εκτιλήσονται αυτή τη στιγμή στο Συμβούλιο. Για τους οργανισμούς ε, εταίρους θα συμφωνήσω και πάλι με την εισηγήτρια θεωρώ βεβαίως ότι χρειάζεται μία ε, αποσαφήνιση των κριτηρίων από πλευράς των κρατών μελών σε σχέση με τον έλεγχο αλλά και την ενιαία κανονιστική ρύθμιση της λειτουργίας αυτών των οργανισμών εταίρων. Είναι απαραίτητη η παρουσία τους, όμως θα πρέπει να ρυθμίσουμε επακριβέστερα τον τρόπο λειτουργίας τους. Αυτές είναι οι γενικές ε, αρχές ε, που διέπουν τις τροπολογίες ε, που θα καταθέσω. Ο στόχος μου είναι να βρω ε, να βρούμε, συγγνώμη, εγκαίρως ε, ικανοποιητικές συμβαστικές λύσεις, να συμφωνήσουμε και με το Συμβούλιο για να συνεχίσει να υπάρχει αυτό το Ταμείο. Ευχαριστούμε. Μάριαν Χάρκιν τώρα και η κυρία Κονέλησαν. Uh, ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την μέχρι τώρα δουλειά της. Ε, προφανώς έχει βάλει σε αυτή την καρδιά της ε, και έχει ακόμα βέβαια και πάρα πολλή δουλειά μπροστά της με όλες αυτές τις ε, τροπολογίες. Κοιτάξτε, στηρίζω πολλά από αυτά που είπατε όπως τις αλυσίδες τροφίμων, τα εθνικά προγράμματα τροφίμων, την αρχή της συνεργασίας να αποφεύγονται... Να αποφεύγουμε να πετάμε τρόφιμα. Όσον αφορά τον προϋπολογισμό, ε, μερικοί ζητάνε την αύξηση. Νομίζω εσείς λέτε ας κρατήσουμε ό,τι έχουμε. Αυτή τη στιγμή γίνονται πάρα πολλές ε, συζητήσεις σχετικά με αυτό. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε κάτι, ίσως μπορείτε να μας ενημερώσετε. Θα με ενδιέφερε να το ακούσω. Ε, εμείς ε, προσπαθήσαμε να πούμε και το εξής, ότι αν κάποια κράτη δεν ε, χρησιμοποιούν χρήματα, μπορούν αυτά να επιστρέψουν στον κοινοτικό προπολογισμό. Ορισμένοι από τους συναντέλφου μου τάσσονται υπέρ της ε, συγχρηματοδότησης και λένε ότι ε, θα πρέπει να προσφερθούν τα χρήματα σε αυτούς που έχουν πραγματική ανάγκη. Βεβαίως ε, η συγχρηματοδότηση έχει και το στοιχείο του πολλαπλασιαστή. Θα δούμε κατά πόσο μπορούμε να επιτύχουμε το συμβασμό. Ένα από τα βασικά πράγματα ε, κατά την άποψή μου, είναι όλη αυτή η διαδικασία εφαρμογής να μην είναι ιδιαίτερα περίπλοκη και πρέπει να εξετάσουμε πολύ προσεκτικά την αξιολόγηση. Πράγματι, Πρέπει να μετρήσουμε το αποτέλεσμα, αλλά ξέρετε ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ότι δεν μπορούμε ε, να στηρίζουμε όλο αυτό το πρόγραμμα σε ΜΚΟ. Χρειαζόμαστε μια, ένα ηχηρό μήνυμα από την Επιτροπή έτσι ώστε να προχωρήσει το Συμβούλιο. Ε, εν πάση περιπτώσει ε, να ξέρουν ότι αυτή, αυτή η Επιτροπή δεν θα σταματήσει να εργάζεται προς τη σωστή κατεύθυνση. Κορνέλισεν και Νομίζω ότι έχουμε περάσει αρκετές ώρες ε, ή έχουμε μπροστά μας ακόμα αρκετές ώρες ευχάριστων ε, συζητήσεων ε, και νομίζω ότι όλα αυτά είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Για μας λοιπόν, για τους πράσινους, υπάρχουν δύο βασικά θέματα. Το ένα είναι ότι τα τρόφιμα που περισσεύουν δεν θα πρέπει να πετιούνται. Η τροπολογία μας 226 ε, ε, στοχεύει ακριβώς αυτό. Και θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτά τα πιστεύει και η κυρία Χάρκιν. Κατόπιν, μην ξεχνάμε, 20 εκατομμύρια τόνοι τροφίμων πετιούνται ε, κάθε χρόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 90 εκατομμύρια συνολικά, αλλά τα 20 εξ αυτών είναι απόλυτα βρόσιμα. Αυτή τη στιγμή ε, γίνεται χρήση των 40.000 τόνων. Ίσως ε, μπορούμε λοιπόν να αποφεύγουμε να πετάμε αυτές τις μεγάλες ποσότητες. Θα θέλαμε στις περίφημες τράπεζες τροφίμων, σε εισαγωγικά βέβαια, να προσφέρουμε όλα αυτά τα τρόφιμα να γίνονται κάποιες ε, συνεννοήσεις ε, με αλυσίδες τροφίμων ε, έτσι ώστε να υπάρχει, να εφαρμοστεί αυτό το πρόγραμμα. Αυτό που θα θέλαμε θα ήταν τελικά πράγματι τα χρήματα να καταλήγουν σε αυτούς που πραγματικά τα χρειάζονται. Κατόπιν τούτου οφείλουμε να δουλεύουμε στοχευμένα. Νομίζω ότι είναι σημαντικό τα κρατη να έχουν τη δυνατότητα ε, να συμμετέχουν, γιατί δεν έχει βέβαια νόημα να τα δίνουμε τα χρήματα αυτά σε κάποια κράτη που ούτε καν τα χρειάζονται, γιατί δεν έχουν τι να τα κάνουν. Και πρέπει βεβαίω και να διαφοροποιήσουμε στη συγχρηματοδότηση τα πλουσιότερα κράτη να πληρώνουν περισσότερο, τα φτωχότερα λιγότερο. Αυτό σημαίνει αλληλεγγύη να υπάρχουν περισσότερα χρήματα. Γιατί αν προβλέπεται η συγχρηματοδότηση για όλους και δεν υπάρχουν αρκετά κονδύλια, καταλαβαίνετε ότι οι χώρες που πραγματικά έχουν ανάγκη ε, δεν βοηθούνται αρκετά. Υπάρχει μία σειρά τροπολογιών που θα ήθελα να ε, αναφέρω σχετικά με την σχετική φτώχεια, να λαμβάνεται υπόψη η σχετική φτώχεια. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτό ισχύει σε αυτή την περίπτωση, γιατί το Ταμείο ασχολείται κυρίως με την ε, ηλική αποστέρηση. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι όταν υπάρχει εξάρτηση διαφόρων κρατών ή οργανώσεων από κοντήλια, αυτό θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Παραδείγματο χάνει στην Ουγγαρία έχουμε περίπου 40.000 ανθρώπους που ε, χρησιμοποιούν τα τρόφιμα από αυτό το ταμείο και αυτό είναι κάτι που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι δεν θα έχουν αυτά τα τρόφιμα από την 1η του 2014 και εφ' εξής. Και υπάρχουν και κάποια άλλα τεχνική φύσεως θέματα που θέλω να επισημάνω. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να βρούμε έναν τρόπο έτσι ώστε η συγχρηματοδότηση να γίνεται από ιδιώτε. Γνωρίζω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι δεν επιθυμούμε τη συγχρηματοδότηση από του ίδιου του οργανισμού βοήθεια. Σωστό αυτό, γιατί θα περιπλέκονται αλλιώ τα πράγματα. Νομίζω όμω ότι θα μπορούσαμε να έχουμε το συγκερασμό ή έτσι ένα μόρφωμα ανάμεσα σε αλυσίδες καταστημάτων ε, και λαχιοφόρους ε, και οργανισμούς που οργανώνουν λαχιοφόρες αγορές. Αυτός είναι ένας καλός ενδιασμός και δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να τον απαγορεύουμε. Για να απλωστευτούν τα πράγματα για τα κράτη-μέλη ε, νομίζω ότι μπορούμε να προάγουμε τους μηχανισμούς σταθερότητας. Και έχω και κάποια ερώτηση προς την εισηγήτρια. Άκουσα ότι είπατε να μην καταβάλλετε πάνω, ένα ποσοστό πάνω από 10%. Ξέρω ότι αυτό ε, ταυτίζεται με κάποιες μεθόδους των περίφημων τραπεζών και των αλυσίδων τροφίμων. Αλλά τι σημαίνει αυτό. Ε, όταν αυτοί ε, μπορούν και συγκεντρώνουν κάποια χρήματα, αυτά τι πρέπει να τα κάνουν. Κυρία Γεζοβιέτσκα, ευχαριστώ. Η πρωτοβουλία σύστασης ταμείου για τους απόρους είναι πολύ σωστή, εύστοχη και απαραίτητη για τον περιορισμό της φτώχειας, που είναι άλλωστε και στόχος της Στρατηγικής Ευρώπη 2020. Χαίρομαι για την ε, μεγάλη δέσμευση της εισηγητρίας και την προσήλωσή της ε, ε, στην έκθεση αυτή που θέλουμε να είναι αποτελεσματική. Θέλω με τις τροπολογίες μου να εξασφαλίσουμε δίκαιη και σωστή αξιοποίηση των κονδυλίων ώστε να αυξήσουμε τον αριθμό των δικαιούχων και να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε το καλύτερο δυνατόν το τομείο. Το 387 προβλέπει δυνατότητα κονδυλίων και κρατικών και τροφίμων που διανέμουν κάποιες φιλανθρωπικές οργανώσεις και επίσης κάποιες εισφορές ή προσφορές μπορούν να γίνουν από διάφορα γραφεία ή καταστήματα. Επίσης, με την τροπολογία 459 μιλούμε για τη δυνατότητα μη επιστροφή ε, του ΦΠΑ. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την ε, οικονομική κρίση και την ε, δυνατότητα να μην μπορέσουν να εκμεταλλευτούν όλοι τα κονδύλια του, τον, του Ταμείου αυτού για τους απόρους, παρόλο που ίσως χρήζουν υποστήριξη. Συμφωνώ με την πρόταση του κυρίου Ορή ότι σημαντικό είναι το θέμα της παρακολούθησης, του monitoring ό,τι αφορά την χρήση αυτών των κονδύλιων, ώστε πραγματικά να πιάσουν τόπο και να φτάσουν στους δικαιούχους. Ε, στην τροπολογία 285 μιλούμε για την προσθήκη επιπλέον δικτών με τον αριθμό των απειλούμενων από τη φτώχεια και των παιδιών. Γιατί νομίζω είναι χαρακτηριστικό και δείκτες ε, για να αποτιμήσουμε την απειλή της στόχης στις ε, διάφορες χώρες μέλη και αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στα πλαίσια της στρατηγικής του 2020. Νομίζω ότι και το Ταμείο για και το Κοινωνικό Ταμείο και ε, το Ταμείο Πόρων είναι σημαντικά, αλλά θα πρέπει να αποφύγουμε επικαλύψεις ε, και γι' αυτό ε, πρότεινα την τροπολογία 242 για να εξασφαλιστεί συντονισμός και όχι επανάληψη των δραστηριοτήτων και επικάλυψη μεταξύ των δύο ταμείων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ την εισηγήτριά μας ε, για τα όσα έχει κάνει, και διότι έχει εργαστεί ήδη σκληρά. Πρωτού περάσω στις λεπτομέρειες των τροπολογιών που κατέθεσα, θα ήθελα να σε επενθυμίσω δύο-τρία σημεία, μεταξύ των οποίων είναι και κάποια σημεία επικαιρότητα θα έλεγα και παραλληλισμού με εργασίες άλλων ε, επιτροπών που συμβάλλουν στις εργασίες μας για την έκθεση της Έμερ Κοστέλο. Αναφέρομαι συγκεκριμένα στην Επιτροπή Γεωργίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης. Αρχίζοντας από την Επιτροπή Γεωργίας, και όπως αντέδρασαν και οι βασικοί ενδιαφερόμενοι φορείς, δηλαδή οι επιστηστικές τράπεζες, Νομίζω ότι οφείλουμε να ε, έχουμε κατά νου μια συνολική εικόνα. Έχουμε την απόφαση του Δικαστήριου της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και ε, την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, μετά από την πάγια και ισχυρή πίεση που ασκεί η δική μας Επιτροπή. Θυμηθείτε και τα ενδιάμεσα στάδια, δηλαδή το προφορικό έτοιμο, προφορική ερώτηση και το καθεξής. Λοιπόν, η Επιτροπή, βασιζόμενη στο άρθρο 175 της Συνθήκης, λαμβάνει δεόντως υπόψη την τελεσίδικη απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι σημαντικό να έχουμε ολόκληρη την εξίσωση στο μυαλό μας, γιατί αν θέλουμε μέσω των τροπολογιών να αποκαταστήσουμε το προηγούμενο πρόγραμμα, δεν θα το πετύχουμε. Η εξίσωση, ξαναλέω, είναι δύσκολη και ο εισηγητής Επιτροπής Γεωργίας ε, κατάλαβε ούτως ή άλλως πως μπορούμε να καταφέρουμε πάρα πολλά. Στο ίδιο πνεύμα που μας προτείνει και η συγκήτρια να καταπολεμήσουμε το θέμα των αποβλήτων τροφίμων, της κατασπατάλησης τροφίμων, των καλών επιστηστικών πρακτικών, αλλά ε, ε, δεν πρόκειται να το πετύχουμε αυτό μέσω ενός ταμείου που απλώς διανέμει τρόφιμα. Μπορούμε όμως να ε, χαράξουμε τον δρόμο και αν υπάρχουν γεωργικά αποθέματα θα πρέπει να επανεισαχθούν μέσα στο μηχανισμό, διότι βασιζόμαστε ούτω ή άλλω σε υφιστάμενα αποθέματα και η νομολογία του δικαστηρίου, δεν μπορεί εν τη αυτή περίπτωση να απαγορεύσει τη χρήση αυτών των αποθεμάτων. Περνώ τώρα στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Ε, θα δούμε ενδελεχέστερα τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώθηκε η επιχειρηματολογία της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης. Μάλιστα, υπήρξε ένας ε, τσακωμός θα έλεγα και κάποιοι το χάρηκαν σε σχέση με τα στοιχεία, τα αριθμητικά που μας έδωσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Σας θυμίζω ότι η αδίποτε τροπολογία σχετίζεται με αριθμητικά στοιχεία του πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου, ούτως ή άλλως θα έπρεπε να κρυθεί μη παραδεκτή. Διότι από την έναρξη των διαπραγματεύσεων και μετά όλοι έλαβαν γνώση της διαφοράς ανάμεσα αφενός στη νομική βάση και αφετέρου ε, στα νούμερα του πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου. Δυνάμεθα να τροποποιήσουμε ε, την πρόταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ε, σε σχέση με το συνολικό ποσό, αλλά σίγουρα δεν μπορούμε εμείς να το κάνουμε ως Επιτροπή Απασχόλησης. Ως εκ τούτου ε, δεν ε, μπορούμε να δεχτούμε αυτές τις τροπολογίες γιατί δεν αναφέρονται στο συνολικό ποσό. Και ξαναλέω ούτως ή άλλως θα έπρεπε να κρυθούν μη παραδεκτές. Υπενθυμίζω ότι πέρα από την πολιτική συμφωνία που επήλθε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ο αγώνας που μας περιμένει θα είναι δύσκολος. Σας υπενθυμίζω δύο στοιχεία προς επίρρωση ε, αυτού του ισχυρισμού. Παρότι στο παρελθόν υπήρχε δημόσια γαλλογερμανική συμφωνία βάσει της οποίας από 1η 2014 θα εξέλιπε αυτό το ταμείο. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ε, στα πλαίσια αυτής της συμφωνίας κινούμεθα και σήμερα. Όμως, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όπου ε, ε, ε πήγανε κάποιοι από εμάς στο Βερολίνο και να παρακολουθήσουν την συζήτηση σε σχέση με την ίδια την ύπαρξη του Ταμείου για τους Απόρους συνειδητοποιούν πόσο κρίσιμη παραμένει η κατάσταση. Έξω και ε, το αίσθημα της συλλογική ευθύνης ε, με το οποίο αντιμετωπίζουμε την, ε, το σχέδιο έκθεσης της ηγήτριάς μας. Αυτά είναι ήδη γενικών σχολείων. Θα περάσω στα ειδικότερα. Για την νομική βάση θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ούτως ώστε ή η πρόταση της Επιτροπής Γεωργίας που ξαναλέω βασίζεται στο άρθρο 175 της συνθήκης να μην αλλάξει και να παραμείνει η βάση ε, αναφοράς χάρη στο οποίο θα λειτουργήσει το Ταμείο για το θέμα της συγχρηματοδότησης, ε, στο οποίο αναφέρθηκαν πολλά μέλη της Επιτροπής. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό το σημείο, πιστεύω, όμως... Ή ε, ελπίζω ότι στην τελική μας θέση θα κατορθώσουμε να συγκεράσουμε διαφορετικές απόψεις. Σε πολλά κράτη-μέλη η κινητοποίηση για την παγκόσμια επιστημιστική ασφαλεία και πιο συγκεκριμένα η βοήθεια προς τους απόρους συνιστά μια πολιτική εκ των ονουκάνευ. Και επανέρχομαι σε αυτά που μας έλεγε η κυρία Σίνκλερ εχθές, ε, μιλώντας για τις δηλώσεις του κυρίου Φανερόμπη για αυτό το θέμα στη στην ανοιχτή διάσκεψη Προέδρων. Για τη συγχρηματοδότηση και επανέρχομαι. Ε, στον μαθηματικό τύπο που θα προτείνουμε τελικά θα πρέπει να επιδείξουμε ευελιξία. Υπάρχουν περιπτώσεις ε, όπου είναι παράλογο να ε, τολμήσουμε να φανταστούμε ή και να προτείνουμε συγχρηματοδότηση διότι πολύ απλά δεν υπάρχουν κονδύλια. Όμως, σε άλλες περιπτώσεις η βοήθεια που θα απορρέει από το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο που θα έχει ε, οικοδομήσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν θα καλύψει ούτε τις ανάγκες αλλά ούτε και τις πρώτερες πρακτικές αυτών των κρατών. Γι' αυτό οι κυβερνήσεις των κρατών, και δεν αποκλείω τη Γαλλία, αποφάσισαν να προσδώσουν πρόσθετη βοήθεια στον μηχανισμό που διαθέτουμε, διότι δεν θα επαρκούσαν τα κονδύλια. Και σε αυτό το πλαίσιο μιλάμε για εθελοντική συνδρομή των κρατών μελών. Ως προς τους όρους διανομής της βοήθειας, θα πρέπει να μεριμνήσουμε ώστε να ανταποκρίνεται στο πνεύμα λειτουργία του Ταμείου. Δεν είναι ε, τεχνοκρατικό, γραφειοκρατικό Ταμείο που απαιτεί ε, τρία διαφορετικά γραφεία ελέγχου, ε, ε, οικονομικού ελέγχου για να ενεργοποιηθεί, διότι ο στόχος είναι να βοηθήσουμε τους απόρους. Ξαναλέω, ο στόχος της Επιτροπής, ο βασικός στόχος της Επιτροπής είναι να καταπολεμήσουμε τον κοινωνικό αποκλεισμό, να ενισχύσουμε την ένταξη των απόρων και γι' αυτό δεν αναφερόμαστε μόνο σε επιστητιστικές τράπεζες και την δωρεάν διανομή, αλλά ε, και των κοινωνικών παντοπολίων, ε, διότι σε αυτό εμπλέκεται μία αγοραστική πράξη που δεν μπορεί να ακυρωθεί μέσω της νομοθεσίας. Υπάρχουν και άλλες σημεία που θα πρέπει να εξακριβώσουμε την συγκεκριά, αλλά οπωσδήποτε θέλω να σχολιάσω μία τροπολογία που κατέθεσα σε σχέση με τη μεταβατική περίοδο. Διότι σήμερα, τη σήμερον ημέρα, Έχω την εντύπωση ότι θα έπρεπε να υιοθετήσουμε ένα μηχανισμό που θα εξασφάλιζε την αίσια του Ταμείου για, την, ε, για το 2014 ο θα επέλθει ε, ρήξη στη λειτουργία του προγράμματος για ένα χρόνο και αυτό θα έχει καταστροφικά αποτελέσματα για τους ενδιαφερόμενους. Η Καρή Μαντελή θα πάρει το λόγο και ο Πατρίκ ρήξη στη συνέχεια. Ευχαριστώ. Δίκαιο έχετε. Έχουμε και τη μεταβατική περίοδο γιατί δεν μας μένει και πολύ χρόνος μέχρι το 2014. Και παρόλο που στη στρατηγική του 2020 έχουμε το στόχο να μειώσουμε μέχρι το 2020 τουλάχιστον τη φτώχεια για 20 εκατομμύρια πολίτες να ξεφύγουν από την εξαθλίωση, δεν ξέρω αν θα προλάβουμε. Και όταν ζητούμε αύξηση του προϋπολογισμού, είναι γιατί ακριβώς υπάρχει τεράστια ζήτηση στην Ευρώπη. Υπάρχει κατακόρυφη αύξηση των αναγκών και ζητούμε ε, αύξηση του προπολογισμού όχι από καπρίτσιο, αλλά γιατί δυστυχώς ε, οι συμπολίτε μας ε, φτωχαίνουν όλο και περισσότερο. Και έχουμε τα κοινωνικά παντοπολία, τις τράπεζες τροφίμων και βρίσκουμε και ένα νέο πρόσωπο. Και με ένα τέτοιο ταμείο που θα έχει ως ε, στόχο ακριβώς τους ε, στέγους και τους απόρους, ε, θα έχουμε πολύ στοχοθετημένη δράση. Δεν μπορούμε να τους πούμε ότι από αύριο δεν θα έχετε πρόσβαση σε τρόφιμα, όταν δηλαδή στερέψουν τα ταμεία. Το θέμα της αύξησης του προπολογισμού είναι επιτακτική ανάγκη λοιπόν. Το δεύτερο που επίσης επισημάνατε εύστοχα είναι το θέμα της απλούστευσης θα πρέπει να μεριμνήσουμε ώστε και η συγκεκριά στην έκθεσή της να απλουστεύσουμε τα πράγματα για να εξασφαλιστεί πρόσκοπτη και άμεση πρόσβαση στο Ταμείο των Δικαιούχων Οργανισμών. Σε ό,τι αφορά τη συγχρηματοδότηση. Εδώ έχω αρκετές απορίες. Μας λέτε ότι υπάρχει το κονδύλιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Δεν θα είναι μια δημοσιονομική γραμμή του Κοινωνικού Ταμείου, αλλά κάτι διαφορετικό. Αλλά θα συστήσουμε αυτό το νέο ταμείο για τους απόρους από ένα τμήμα του συνολικού κονδυλίου, του συνολικού προϋπολογισμού του ΕΚΤ, αν, κάνω, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή παίρνουμε κονδύλιο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, μια μεταφορά ουσιαστικά κονδυλίου από το ΕΚΤ στο, στο Ταμείο Αστέγων στο Ταμείο Απόρων, συγγνώμη. Συγγνώμη που σα διακόπτω, αλλά θέλω να το διευκρινίσω. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στήριξε την πρότασή τη στο άρθρο 175 παράγραφο 3. Το άρθρο 175 παράγραφο 3 τη συνθήκη περιλαμβάνεται στο, στο κεφάλαιο 18 της συνθήκης που αφορά την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή. Και η παράγραφος 3 προβλέπει αν χρειαστούν ειδικέ δράσεις στα πλαίσια του Ταμείου υπό την επιφύλαξη των μέτρων άλλων πολιτικών της Ένωσης, οι δράσεις αυτές μπορούν να εγκριθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το καθεξής. Και τα εν κονδύλια αναφέρονται στο παράγραφο 1. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, θα στηρίξει με τις δράσεις της ε, την πραγμάτωση αυτών των στόχων με κάποια διαρθρωτικά κονδύλια. Ε, ΦΕΟΓΑ, Τμήμα Προσανατολισμού, ε, Κοινωνικό Ταμείο και Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Πρόκειται λοιπόν για το σύνολο των διαρθρωτικών ταμείων που αναφέρονται στο άρθρο. Δεν ε, μιλούμε μόνο για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Είναι σημαντικό να έχουμε αυτό υπόψη, δηλαδή τι ακριβώς σημαίνει η μνήα της Ευρωπαϊκής Επιτροπή, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της Νομικής Βάσης του άρθρου 175, παράγραφος 3. Αυτό ας μην το λησμονούμε. Ναι, ναι, αλλά τώρα δεν καταλαβαίνω τι ισχύει. Αν λέτε ότι πρόκειται για το συνολικό προϋπολογισμό των διαστατικών ταμείων, τότε Α, τι γίνεται όταν θα δημιουργήσουμε το νέο ταμείο. Θα υπάρξει μια μεταφορά γιατί για τα διαρθρωτικά ταμεία ισχύει 50-50. Αν μου πείτε ότι μιλούμε για το συνολικό κονδύλιο, τότε ε, είναι τμήμα των διαρθρωτικών ταμείων. Οπότε μπορούμε να εφαρμόσουμε και το μοντέλο 80% και 95% για την Ελλάδα. Διαρωτώ με όμως, οι χώρες που αντιμετωπίζουν δημοσιονομικές δυσκολίες, πώς θα εξασφαλίσουν ε, το ποσοστό της χρηματοδότησης για να μπορέσουν να αξιοποιήσουν τα κονδύλια του Ταμείου. Δεν θα πρέπει σε περίοδους κρίσης χώρες όπως η Κύπρος, η Ελλάδα ε, να διευκολυθούν. Αν δεν μπορούν να εξασφαλίσουν ε, το, τη συγχρηματοδότηση, ακόμη και είναι αυτή μόνο 5%. Γιατί αν τους λείπει το 5% δεν θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν το 95% ενώ ε, ο δικός τους πληθυσμός είναι αυτός που κατεξοχή έχει ανάγκη αυτά τα κονδύλια. Έχουμε την γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης ε, που ε, προτείνει διάφορα σημεία για την ενίσχυση της έκθεσης. Καταρχήν η ποιότητα των τροφίμων. Το είπα και στην Επιτροπή. Είναι σκανδαλώδες ε, να ακούμε για σκάνδαλα επισητιστικά και να περιμένουμε το σκάνδαλο του αλογίσιου κρέατος και να λέμε «Α, πόσα τρόφιμα πάνε χαμένα, ας τα δώσουμε στους απόρους» και οι άποροι δικαιούνται υγιή και ποιοτικά τρόφιμα. Όχι μόνο τα σκάρτα. Είναι σημαντικό λοιπόν το θέμα της ποιότητας και της υγείας των τροφίμων. Πρόθεση της κοινωνικής καινοτομίας. Εκεί που θα πρέπει να βοηθήσουμε ώστε να δημιουργηθούν κοινωνικά παντοπολία. Γιατί ενισχύεται η αλληλεγγύη στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας. Γιατί ενισχύονται οι κοινωνικοί δεσμοί, ενισχύεται η κοινωνική οικονομία. Είναι ευάρεστος αυτός ο στόχος και θα πρέπει ε, να το τονίσουμε στην έκθεσή μας. Ε, είμαι και οικολόγος. Θα πρέπει να καταπολεμήσουμε την κατασπατάληση και η λύση είναι μία, αλλαγή του μοντέλου. Και στο νέο μοντέλο θα πρέπει να ενισχύσουμε το θέμα της αξιοποίησης των ε, βραχίβιων αλυσίδων και κυκλωμάτων παραγωγής και διανομής τροφίμων. Έτσι θα αναπτύξουμε και ε, την τοπική οικονομία, αλλά θα ενισχύσουμε και το αίσθημα της, τοπικής αλληλεγγύης. Αυτά, κυρία Πρόεδρε, και περιμένω με ανυπομονησία τις συμβαστικές προτάσεις, αλλά και γενικώ ε, την τελική διαμόρφωση της έκθεσης. Ευχαριστώ, Πατρίκ Λιαρίκ. Και μετά η Ελισαμπέθ Σρέντερ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την κυρία Κοστέλο για την προσπάθειά της και να σας ευχαριστήσω και εσάς κυρία Πρόεδρε για τις διευκρινήσεις που μας κάνατε. Θα πρέπει να έχουμε επίγνωση ότι το έργο που επιτελούμε εδώ ε, είναι πολύ σημαντικό και το περιμένουν πώς και πώς οι συμπολίτες μας παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν δημιουργηθεί ψηλές προσδοκίες. Θα ήθελα να επισημάνω μερικά προβλήματα. Ε, παρά τις διευκρινήσεις που μας δώσατε κυρία Πρόεδρε, δεν είμαι βέβαιος ότι το νομικό καθεστώς ε, αυτής της πρότασης ε, στα πλαίσια του άρθρου που αναφέρατε ως νομική βάση, το 175 δηλαδή παράγραφος 3, ε, είναι δεδομένο. Οπότε σκόπιμο και χρήσιμο θα ήταν είτε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή από την Νομική Υπηρεσία να δοθούν κάποιες διαβεβαιώσεις και χέγγια για το θέμα αυτό. Επίσης, ένα συναφές ζήτημα. Πώς θα χρηματοδοτηθεί αυτό το νέο ταμείο. Θα γίνει μια απλή μεταφορά κονδυλίων ή διαφορετική κατανομή των κονδυλίων εντός του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Δεύτερη παρατήρηση. Αντιλαμβάνομαι ότι δεν μπορούμε εδώ να δώσουμε μάχη για συγκεκριμένα ποσά. Απ' την άλλη, δεν μπορούμε να μένουμε ε, χωρίς κανένα ποσό, χωρίς κανένα αριθμό, ε, σε γενικότητες και αφησιμίες, γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέρριψε το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, ενώ για συγκεκριμένες δράσεις ε, εμείς δεν θα προτείνουμε κανένα ποσό ή θα δεχτούμε περικοπές ή μείωση. Γιατί ουσιαστικά μείωση προτείνεται μέχρι τώρα, ούτε καν στα σταθερότητα. Υπάρχει λοιπόν και μεταξύ μας μία ασυνέπεια και θα πρέπει να το προσέξουμε αυτό. Δεν μπορούμε να αφήνουμε τέτοια βεβαιότητα να πλανάται στην ατμόσφαιρα. Γιατί οι οργανώσει έχουν συγκεκριμένα ποσά. Τόσα συσίτια, τόσα γεύματα προσφέρουν το χρόνο, ε, τόσο κοστίζουν. Θα πρέπει να μπορούν και αυτέ οι οργανώσει να κάνουν μια μακροπρόθεσμη πρόβλεψη των δράσεών του και του προπολογισμού του. Παρόλο που αντιλαμβάνομαι το επιχείρημά σα ότι δεν μπορούμε να έχουμε συγκεκριμένα ποσά. Επίση επικαλούμαστε τη στρατηγική του 2020 με το στόχο τη μείωση ε, κατά 20 εκατομμύρια, των φτωχών τη Ευρωπαϊκής εγώ ούτε λέξη δεν πιστεύω από όλα αυτά. Θεωρώ ότι είναι ε, ανέντιμες ε, φλιαρίες ε, και αρλούμπες ουσιαστικά που παρουσιάζουμε στον κόσμο. Δεν πρόκειται να μειωθεί ο αριθμός των φτωχών, αντίθετα θα αυξηθούν οι φτωχοί εργαζόμενοι Έχουμε γυναίκες που μένουν μόνες τους, ε, εργάζονται και παρόλα αυτά χρειάζεται να πάνε στα κοινωνικά συσίτια ή να προσφύγουν στις ε, τράπεζες τροφίμων. Είναι πραγματικά απαράδεκτο και δεν νομίζω θα βελτιωθεί η κατάσταση όπως πάμε. Ναι βέβαια, ναι με θα πρέπει να καταβάλουμε προσπάθεια για να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας, να γίνουν λιγότερο επισφαλείς θέσεις απασχόλησης, να αναβαθμιστεί η ποιότητα αλλά δεν οδεύουμε προς αυτό το δρόμο, γιατί κάθε εβδομάδα όλο και πιο αρνητικές ε, πληροφορίες και ζωφερή εικόνα ε, λαμβάνουμε. Ε, κάτι άλλο για το οποίο συμφωνούμε όλοι, αλλά θα ήθελα να το επαναλάβουμε και να το διατρανώσουμε. Έχουμε και μία σημαντική διοικητική περιπλοκή στην πρόταση. Θα πρέπει να απλουστεύσουμε τις διοικητικές διατυπώσεις Αλλιώς θα χρειαστούμε εμπειρογνώμονες, λογιστές, ε, νομικούς και τους οποίους θα πρέπει να πληρώνουμε αδρά για να μας διευκρινίζουν την κατάσταση. Και τέλος, αν βρούμε ένα σύστημα το οποίο εμείς θα πρέπει να επινοήσουμε για να αποφύγουμε αυτή την κατασπατάληση των τροφίμων και να μπορέσουμε σε συνεργασία με τους παραγωγούς αλλά και με το, τις αλυσίδες διανομής να μπορέσουμε αυτά τα τρόφιμα αντί να τα πετάμε και να τα σπαταλάμε να τα δώσουμε σε φιλανθρωπικές οργανώσεις για να αξιοποιηθούν για ευαγείς σκοπούς. Επίσης δεν έχουμε μόνο το θέμα των τροφίμων εδώ, δεν είναι μόνο το επιστηστικό ζήτημα το δεχόμαστε και ζητούμε αύξηση του προπολογισμού γι' αυτό, αλλά ταυτόχρονα ας μην ξεχνούμε και το θέμα της επισητιστικής βοήθειας. Γιατί αλλιώς ε, θα επιδεινωθεί η καθημερινότητα πολλών συμπολιτών μας δυστυχώς. Ευχαριστώ. Η Ελιζαμπέτ Σρέτερ και μετά η κυρία Μωράν Σάχτιε. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ ε, θα ήθελα απλά να στηρίξω τον κύριο Ρή και την κυρία Χάρκιν όσον αφορά το θέμα του εθελοντισμού ε, και του προαιρετικού στοιχείου. Δηλαδή μπορούν να συμμετέχουν μόνο αυτά τα κράτη που το επιθυμούν και που δεν έχουν διαφορετικό σύστημα. Όλα τα άλλα δεν έχουν νόημα γιατί γνωρίζουμε ότι αυτά έχουν άμεση σχέση ε, και προσμετρώνται στα κονδύλια του κράτους μέλους σε σχέση με το Ταμείο Σταθερότητας. Δηλαδή, αν ένα κράτος μέλος επιθυμεί να εφαρμόσει άλλα προγράμματα από, που έχουν σχέση με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για την ε, φτώχεια και παράλληλα θέλει να εφαρμόσει και ένα λειτουργικό πρόγραμμα, υπάρχει μια σειρά κρατών μελών τα οποία έχουν τα δικά τους ε, τα ε, τοπικά προγράμματα για τα κοινωνικά παντοπολία. Έχουν βρει δηλαδή τα κράτη αυτά άλλους ε, μηχανισμούς και κατόπιν τούτου όλα αυτά που λέμε εμείς δεν βοηθούν. Ξέρουμε ότι μέχρι τώρα υπάρχουν 19 κράτη που έχουν καταφύγει σε αυτή τη βοήθεια. Έχουμε λοιπόν κράτη όπως η Γερμανία και η Μεγάλη Βρετανία. Αν έπρεπε τα κράτη αυτά να καταφύγουν σε αυτό το ταμείο, τότε δεν θα έμενε τίποτα άλλο για τα υπόλοιπα κράτη. Γιατί η Γερμανία είναι μια τεράστια χώρα, ε, ε, χαρακτηρίζεται από πολύ μεγάλη φτώχεια, αν και θεωρείται πλούσια. Για μας λοιπόν έχουμε υπολογίσει ότι αν η Γερμανία κατέφευγε θα χρειαζόταν τουλάχιστον 500 εκατομμύρια αν βέβαια εφαρμόσουμε τα κριτήρια που προτείνει η Κομισιόν. Η Γερμανία όμως έχει το δικό της το εθνικό σύστημα για τα συσίτια, συγγνώμη, για τα κοινωνικά παντοπολία και τα συσίτια. Ε, και αυτά λειτουργούν πολύ καλά ε, είναι συστήματα που δεν θέλουμε να τα καταστρέψουμε, δεν θέλουμε ξαφνικά να επιβάλλουμε κοινοτικά συστήματα τη στιγμή που επιτόπου ισχύουν πάρα πολύ καλά τέτοιου είδου ε, συστήματα βοήθειας και αλληλεγγύη. Μέχρι τώρα έχουμε 19 κράτη που εξαρτώνται από ε, το δικό μας, το μεταβατικό σύστημα. Όπως σας είπα υπάρχουν ε, άλλα κράτη για τα οποία ισχύουν τελείως διαφορετικές καταστάσεις. Γι' αυτό λοιπόν το προαιρετικό στοιχείο το βρίσκω καθοριστική σημασίας. Το δεύτερο που θέλω να πω ε, και το λέω γιατί δεν είπε τίποτα επ' αυτού η εισηγήτρια. Υπάρχουν τροπολογίες ε, που καταργούν την αξιολόγηση, που καταργούν την έγκριση λειτουργικών προγραμμάτων και εγώ επειδή ασχολούμαι με τα διαφορετικά ταμεία εδώ και πάρα πολύ καιρό θεωρώ ότι κάτι τέτοιο είναι ανεύθυνο. Είναι ανεύθυνο εφόσον ενδιαφερόμαστε για τα χρήματα του Ευρωπαίου Φορολογούμενου. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να υπάρχουν ελάχιστοι έστω κανόνες, όπως ισχύουν και αλλού και για αυτά τα ταμεία. Ε, θα ήθελα βέβαια ε, να μας πει η τι πιστεύει για αυτές τις ε, τροπολογίες. Κατόπιν αναφέρθηκε ότι για τα προβλήματα που μαστίζονται από την κρίση υπάρχει πρόβλημα γιατί δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τη συγχρηματοδότηση. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια πρόταση, πρόκειται για ένα μηχανισμό ο οποίος υπάρχει και στα διαρθρωτικά ταμεία, μόνο που ε, υπάρχουν πολλές τροπολογίες διαγραφής σχετικά με το μηχανισμό αυτό. Και όλα αυτά απορρέουν από το ότι ε, παίζουν και άλλα μακροοικονομικά στοιχεία. Κοιτάξτε, εγώ δεν έχει νόημα να διαγράψουμε αυτό τον μηχανισμό επειδή υποτίθεται αυτός ε, ε, αντιτίθεται σε μακροοικονομικές εξελίξεις. Ακριβώς για αυτό το λόγο πρέπει να υπάρχει ο μηχανισμός και θα με ενδιαφέρε ε, να ακούσω τι λέει η συγκήτρια από αυτού. Όσον αφορά τον περιορισμό των μέσων, κοιτάξτε, στην επίσημη δημοσιονομική πολιτική ε, χρειαζόμαστε αριθμούς, χρειαζόμαστε στοιχεία. Δεν μπορούμε να λέμε επειδή χρειαζόμαστε περισσότερα κονδύλια παραμένει το ποσό ανοιχτό. Ε, η ευθύνη μας είναι να χειριζόμαστε υπεύθυνα τα χρήματα των φορολογουμένων και έστω και με τα λίγα κονδύλια που έχουμε, πρέπει να τα χρησιμοποιούμε και αυτά κατά τον βέλτιστο δυνατό τρόπο. Αυτή λοιπόν η συζήτηση που πρέπει να διεξάγουμε. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την νομική βάση. Πρώτα όμω την κυρία Μωρά Σάτχε. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι πρώτα απ' όλα θα πρέπει να συμφωνήσουμε ως προς ότι η αξία τη αλληλεγγύη είναι από τι θεμελιώδει αξίε και ιδρυτικέ αξίε τη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως είπε η κυρία Σρέντερ, και σε εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, το θέμα της αλληλεγγύης είναι ένα ζήτημα και άσχετα με τα μέτρα που θα εγκρίνουμε, η αλληλεγγύη θα πρέπει να διέπει όλες μας τις δράσεις. Άλλωστε σήμερα περισσότερο από ποτέ είναι απαραίτητη για εκατομμύρια ανθρώπους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το δεύτερο είναι ότι δεν έχουμε στατιστικά στοιχεία. Διερωτώ με λοιπόν, μήπως δεν βολεύει και όλα μερικούς και στην Ένωση και στα κράτη-μέλη το γεγονός αυτό, γιατί οι ανάγκες συνεχώς αυξάνονται. Την περασμένη Παρασκευή είχα συνάντηση με φιλανθρωπικές οργανώσεις και μου είπαν ότι στην Ήπεθρο πάνω από το 30% των συσιτίων, πάνω από το 30% των ε, είναι η αύξηση στην Ήπεθρο. Βλέπετε λοιπόν ότι μια τέτοια αύξηση στην ανάγκη των συσιτίων είναι ανατριχιαστική και πραγματικά ε, δεν θα είχα καταλάβει τις διαστάσεις του προβλήματος αν δεν μου έλεγαν 30% αύξηση φέτος στα συσίτια. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα ενισχύσουμε αυτό το ταμείο ώστε να εφαρμόσουμε εμπράκτος την αλληλεγγύη και για να τα καταφέρουμε θα πρέπει να συγκεντρώσουμε ακριβή στατιστικά στοιχεία. Είναι πολύ λεπτή η κατάσταση. Έχω καταθέσει σχετικές τροπολογίες και ξέρω ότι οι φιλανθρωπικές οργανώσεις λένε ότι ε, με τη νέα πρόταση αυξάνεται το γραφειοκρατικό άχθος κτλ. Αλλά θα πρέπει και οι χώρες να ενταχθούν στη διαδικασία αυτή. Επίσης, το Ταμείο αυτό για την ε, συνδρομή των ε, απόρων τροποποιεί τη συνέχεια ως προς την εμβέλειά του. Ε, είπαν ο κύριος Σολή και η κυρία Σρέντερ ότι σε τελική ανάλυση τα κράτη-μέλη που δεν θεωρούν ότι χρειάζονται κάτι τέτοιο γιατί έχουν άλλου είδους οργανώσεις. Το θέμα είναι ότι έχουμε όλο και περισσότερους νέους σήμερα. Τα κοινωνικά παντοπολία ε, αρχίζουν και εμφανίζονται ακόμη και στα πανεπιστήμια και αυτό πραγματικά κρούει τον κόδωνα του κινδύνου και αποδεικνύει ότι η κρίση αυξάνεται και αυξάνει και τον αριθμό των ε, ε, απόρων που έχουν τέτοιες ανάγκες. Οπότε θα, είναι λογικό να αλλάζει η εμβέλεια. Αλλά να μην ξεχνούμε ότι η μάχη που δίνουμε για τα ποσά δεν είναι αυτός σκοπός έχει κάποιο νόημα. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες, να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες και δεν μπορούμε ταυτόχρονα να μειώνουμε κατά ένα δισεκατομμύριο τα διαθέσιμα κονδύλια ενώ ταυτόχρονα αυξάνουμε ε, τις ανάγκες του Ταμείου διαπαιδαγώγηση, παιδεία, διαιτολογία, ναι, με τα τρόφιμα και τα επιστημικά θέματα είναι ο πρωταρχικός σκοπός, αλλά βλέπω ότι αυξάνονται και άλλες ε, διαστάσεις, άλλες πτυχές του Ταμείου. Εγώ θεωρώ ότι η μάχη για τα νούμερα δεν θα πρέπει να είναι πολιτική αντιπαράθεση, αλλά θα πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας γιατί καλούμαστε να προασπίσουμε την ίδια την ουσία, την πεπτουσία του Ταμείου. Με τον Φίλιπ Πουλό θα υποβάλουμε προτάσεις για μέτρα πλούστευσης, γιατί θα πρέπει να πλουστευτεί η πρόσβαση στο Ταμείο. Είναι θεμελιώδης προϋπόθεση προκειμένου να υλοποιήσουμε το σκοπό του Ταμείου και να ανταποκριθούμε στις ανάγκες. Και ευχαριστώ την κυρία Κωστέλα, την που θα λάβει υπόψη παρατηρήσεις. Πριν δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα ήθελα να σα υπενθυμίσω ότι για το θέμα των ποσών των αριθμών δεν χρειάζεται να κάνουμε πολιτικά κηρύγματα εδώ και να δίνουμε μαθήματα. Και σίγουρα αν κληθούμε να αποφαθούμε για το θέμα αυτό θα επαναφέρουμε το κονδύλι στο παλιό πρόγραμμα. Και σίγουρα δεν θα δεχτούμε τη μείωση του 40% που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οπότε οι μικροκομματικές παρατηρήσεις που κάνουν μερικοί πέραν των κανόνων που ισχύει την Επιτροπή μας νομίζω ότι είναι απαράδεκτες στα πλαίσια της συζήτησης στην Επιτροπή. Δεν θα πρέπει να γίνεται τέτοια μικροκομματική χειραγώγηση του θέματος των ποσών. Κυρία Ντελάγκερ, μετά τη συζήτηση που έγινε Θέλετε να μας διευκρινίσετε την ε, προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη νομική βάση, που, το άρθρο που επιλέξετε ως νομική βάση για την πρόταση. Yes, I will start with precisely... Ε, ε, Θα αρχίσω ακριβώς με αυτό το σημείο. Το Ταμείο που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι μέσω της κοινωνικής συνοχής και άρα υπάγεται στο άρθρο 175 δάφιο 3 της συνθήκες απευθύνεται στις πληθυσμιακές ομάδες που έχουν αποκλειστεί σε τόσο μεγάλο βαθμό και τόσο απέχουν από την αγορά εργασίας που δεν καλύπτονται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Ο στόχος να καλυφθεί ένα κενό δηλαδή στην πολιτική συνοχή μας. Ο λόγος ε, για τον οποίο εισηγηθήκαμε ένα ταμείο που να κρα... λείπτει όλα τα κράτη-μέλη και είναι υποχρεωτικό. Είναι διότι θέλουμε να καλυφθούν ακριβώς οι πλέον άποροι. Για τα συνοδευτικά μέτρα, ο συνδυασμός ε, ε, των τροφίμων, των επιστημιστικών με άλλων υλικών αναγκών και τις δραστηριότητες που προτείνουμε για να συμπεριληφθούν αυτές οι πληθυσμιακές ομάδες στην κοινωνία είναι στον πυρήνα της πρότασης ε, διότι η δωρεάν διανομή είναι το σημείο εισόδου για να πλησιάσουμε αυτούς τους ανθρώπους ε, που είναι άποροι για να τους βοηθήσουμε να ξεφύγουν από τη φτώχεια. Ο, για την απλούστευση, ε, φυσικά αυτό το Ταμείο εντάσσεται στην πολιτική κοινωνικής ε, συνοχής ε, και άρα εξυπηρετούνται οι στόχοι της κοινωνικής ε, συνοχής, μεταξύ των οποίων και η μεικτή διαχείριση. Αντιλαμβανόμαστε ότι αυτοί οι κανόνες δεν είναι οι ευχερέστεροι και απλούστεροι προς την υλοποίηση και γι' αυτό είναι μάλλον μακρύς ο κανονισμός. Προσπαθήσαμε όμως να ε, βελτιώσουμε και να πλουστεύσουμε την κατάσταση όπου ήταν αυτό δυνατό ε, για τις ε, προκαταβολές, για την μέθοδο υπολογισμού του κόστους, για να προσαρμοστούμε ακόμη και στους οικονομικούς ελέγχους με τους κανονισμούς των ταμείων, παρότι πρόκειται για απόρους. Θα... Η διαχείριση του Ταμείου αναλαμβάνεται από τις ε, ε, διαχειριστικές ε, εθνικές αρχές που ασχολούνται και με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο με στόχο πάλι την απλούστευση στην υλοποίηση των διατάξεων και φυσικά προβλέπεται ότι θα λειτουργήσει αυτή η διάταξη στην πράξη. Για τη συγγραμματοδότηση να κάνω ένα τελευταίο σχόλιο. είναι μια βασική αρχή της μεικτής διαχείρισης και των αρχών της πολιτικής συνοχής. Αφενός ε, θα ε, επιφέρει επιπρόσθετους πόρους στο Ταμείο και αφετέρου ε, για κράτη που έχουν δημοσιονομικούς περιορισμούς με τις προσαυξήσεις ε, τα ε, περίφημα top-up θα φτάσουν στο 95% ε, για τη συγχρηματοδότηση. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, κυρίως για την προχρηματοδότηση της τάξης του 11%, διευκολύνοντας έτσι τη διαχείριση ρευστότητας των κρατών μελών και αυτό το 11% όντως επιτρέπει να χρηματοδοτηθεί πλήρως το πρώτο έτος υλοποίησης έτσι, τα κράτη-μέλη μπορούν να, λάβουν τα, να ανακτήσουν τα ποσά προτού εκινήσει το επόμενο έτος χρηματοδότηση. Θα σταματήσω εδώ. Ευχαριστούμε η συγγήτριά μας. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και πάλι όλα ε, τα κρατημέλη για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Σίγουρα υπάρχουν ε, πολλά στοιχεία κοινά για όλους μας, ε, αλλά υπάρχουν και αρκετά θέματα που διαφωνούμε, γιατί όπως ξέρουμε ο... στη λεπτομέρεια βρίσκεται ο διάβολος και θα πρέπει να καταλήξουμε σε κάποιες συμβαστικές προτάσεις. Αυτά λοιπόν τα κοινά θέματα που μας ενώνουν όπως είπα και προηγουμένως, έχουν σχέση με τις απλουστευμένες διαδικασίες. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι όλοι όσοι μίλησαν σήμερα μίλησαν για το τι είναι απαραίτητο να υπάρξει απλούστευση και παράλληλα, όπως είπε και η κυρία Σχόντα, να αναγνωρίσουμε ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει αξιολόγηση αλλά και λογοδοσία. Είπα ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει απλούστευση των διαδικασιών και αξιολόγηση. Τα ανέφερα αυτά. Νομίζω όμως ε, ότι ε, πρέπει τελικά να δούμε τις τροπολογίες και να δούμε πώς θα μπορέσουμε να ε, επιτύχουμε βελτίωση ως προς τις διαδικασίες. Όλοι όσοι μίλησαν ανέφεραν ότι το Ταμείο αυτό υποσύσταση αφορά τους ε, πραγματικά άπορους και πολλοί αναφέρθηκαν στην στρατηγική 2020. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση 43 εκατομμύρια ανθρώπους ε, που ζουν ε, σε συνθήκες φτώχειας και επίση πάρα πολλούς άλλους που κινδυνεύουν να κατρακυλήσουν στη φτώχεια. 20.000 άνθρωποι δεν καλύπτονται και Βεβαίως το ταμείο αυτό δεν είναι απαραίτητα ένα ταμείο το οποίο θα ασχολείται με την καταπολέμηση της φτώχειας, ασχολείται περισσότερο με το να καλύπτει τις βασικές ανάγκες των ανθρώπων και όπως είπε και η Επιτροπή ε, θα πρέπει να ε, υπάρχει η δυνατότητα πρόσβαση στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και στις υπηρεσίες που προσφέρει το πρόγραμμα. Κατόπιν το θέμα της ε, συγχρηματοδότησης και αυτό προκάλεσε σήμερα πολλές αντιδράσεις. Νομίζω ότι πράγματι υπάρχουν κοινά στοιχεία για αυτό, αλλά υπάρχουν και άλλοι τομείς όπου πρέπει να ορίσουμε πώς θα λειτουργήσουν αυτά στην πράξη. Μεγάλες ανησυχίες υπάρχουν για το ότι κυρίως χώρες που αυτή τη στιγμή καλύπτονται από προγράμματα ότι κάποια κρατημέλη δεν θα μπορέσουν να προσφέρουν την συγχρηματοδότηση και από εκεί θα εξαρτηθεί κατά πόσον θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ή όχι. Εμείς όμως έχουμε στόχο να άρουμε τα εμπόδια για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα. Ε, πολλοί επισήμαναν το θέμα της προαιρετικής συγχρηματοδότησης, της ιδιωτικής συγχρηματοδότησης αυτά ε, είναι σκέψεις που πράγματι αξίζουμε να ασχοληθούμε με αυτές, ίσως με περισσότερες λεπτομέρειες. Κατόπιν, όσον αφορά τους δείκτες και την ε, κλίδα κατανομής ε, και αυτά προκάλεσαν αρκετές αντιδράσεις για το πώς ακριβώς θα λειτουργήσει η κλίδα κατανομής, όπως και οι δείκτες. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι είναι σημαντικό οι δείκτες που χρησιμοποιούμε να είναι σταθεροί και να διασφαλίζουν ότι οι πραγματικά άποροι αυτοί να μπορούν να έχουν πρόσβαση στο πρόγραμμα και ότι το πρόγραμμα θα χρηματοδοτεί τις χώρες εκείνες που έχουν πραγματικά ανάγκη. Αυτός εξάλλου είναι ο στόχος και όλων μας. Πράγματι υπάρχουν κάποιες τροπολογίες όπως αυτές που ε, προέρχονται από την Επιτροπή Γεωργίας και έχουν σχέση ε, με τα παρεμβατικά αποθέματα. Αρκετοί αναφέρθηκαν σε τροπολογίες που προέρχονται από αυτή την Επιτροπή. Έχω την εντύπωση ότι τα αποθέματα ε, από, τα παρεμβατικά, από την παρέμβαση θα πρέπει και αυτά να προσφέρονται, να διατίθενται. Ως προς την ε, συγχρηματοδότηση, το πρόγραμμα MDP, όπως υπάρχει αυτή τη στιγμή, δεν προβλέπει την δυνατότητα συγχρηματοδότησης. Άρα αξίζει τον κόπο να τη σκεφτούμε και εδώ τη συγχρηματοδότηση. Το θέμα της ε, προαιρετικής συμμετοχής. Γι' αυτό θα υπάρξουν πολλές συζητήσεις. Όπως είπε και η Επιτροπή, το Ταμείο έχει ως στόχο τους πραγματικά άπορους σε όλες τις χώρες, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που ζουν σε ακραίες συνθήκες φτώχειας, στερούνται τα πάντα σε όλες τις χώρες. Εγώ προσωπικά επισκέφθηκα μια τράπεζα τροφίμων στο Μάντσεστερ Ξέρω ότι υπάρχουν πολλές οργανώσεις στο ΕΒ Βασίλειο που διαμαρτύρονται ότι δεν τους προσφέρεται το πρόγραμμα και αν ε, μπορούσαν να συμμετέχουν θα μπορούσαν να αποκτήσουν και άλλα κονδύλια αλλά χωρίς τη ρήτρα της ε, συγχρηματοδότησης. Το πρόγραμμα ως ε, έχει προσφέρει μόχλευση, προσφέρει περισσότερα κονδύλια στις οργανώσεις που συμμετέχουν. Η κυρία Κορνέλσεν ε, έκανε ένα ερώτημα σχετικά με τις ε, τροπολογίες που σχετίζονται με την ε, δυνατότητα να χρεώνονται κάποια χρήματα για τα τρόφιμα που προσφέρονται Βέβαια ε, τροποποίησε και πάλι την ε, τροπολογία της αυτή και είπε ίσως ένα είδος συνεισφοράς. Αν μπορούμε να προβλέψουμε ότι ποια χρήματα που στρέφονται θα επιστρέφονται στους ε, αρμόδιους οργανισμούς, γιατί ας μην ξεχνάμε, εδώ μιλάμε για πολύ μικρά ποσοστά και να μην ξεχνάμε ότι ο πραγματικός στόχος τελικά δεν είναι να συγκεντρωθούν χρήματα, αλλά να διασφαλίσουμε την αξιοπρέπεια των τελικών αποδεκτών, να μην στιγματίζονται οι άποροι αυτοί, να μην αισθάνονται ότι ε, λαμβάνουν ελεημοσύνη. Να νιώθουν και αυτοί ότι κάτι συνεισφέρουν στο ταμείο. Αυτό βέβαια πρέπει να το εξετάσουμε. Και νομίζω ότι κατά τη διάρκεια των επόμενων ε, συνεδριάσεων μπορούμε να το δούμε το θέμα. Όσον αφορά τώρα στον προπολογισμό, όπως και όλοι οι άλλοι, και εγώ συμφωνώ ότι ε, δεν φτάνουν τα κονδύλια, ε, όπως είπε και η Πρόεδρος. Βέβαια, η άποψή μας είναι ότι ο προϋπολογισμός πράγματι δεν αρκεί και μπορούμε ε, να προσπαθήσουμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει ως Κοινοβούλιο να επηρεάσουμε αυτά που διαδραματίζονται στο Συμβούλιο σε σχέση με τον προϋπολογισμό αλλά και με τη νομοθετική πρόταση. Δεν έχουμε το περιθώριο να τροποποιήσουμε τον προϋπολογισμό. Νομίζω η κυρία Χάρκιν έκανε μία ερώτηση σχετικά με την πρόοδο στο Συμβούλιο. Και από ό,τι κατάλαβα, οι συζητήσεις που συνεχίζονται σε επίπεδο Συμβουλίου είναι ουσιαστικές, αναμφίβολα, υπάρχει αντίδραση στο πρόγραμμα αυτό και που δεν είναι σαφές ότι σε επίπεδο Συμβουλίου τελικά θα υπάρξει συμφωνία. Συμφωνώ με αυτούς που μίλησαν ότι είναι σημαντικό η Επιτροπή αυτή αλλά και το Κοινοβούλιο να εκπέμψουν ηχηρό μήνυμα υπέρ αυτού του προγράμματος και ό,τι και αν κάνουμε να το κάνουμε για να ενισχύσουμε την πρόταση να διασφαλίσουμε ότι επουδενή δεν θα τεθεί σε κίνδυνο η νομική βάση ε, πάνω στην οποία βασίζεται το πρόγραμμα. Ευχαριστώ την Κομισιόν για τη συνεργασία όσον αφορά την πρόταση και το ότι ε, προσφέρθηκαν να απαντήσουν ερωτήσεις, να συνεργαστούν με μένα, με τους ε, συνεργάτες μου. Εκτιμώ ιδιαίτερα το γεγονός ότι η Κομισιόν ε, παραμένει προσιλωμένη στην ιδέα των απλουστευμένων διαδικασιών και παράλληλα πιστεύω ότι τα μέλη αισθάνονται ότι υπάρχει ένα πολύ ευρύτερο περιθώριο για περαιτέρω απλούστευση και παράλληλα όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, αναγνωρίζουν ότι είναι απαραίτητο να διασφαλίσουμε την ύπαρξη στατιστικών δεδομένων, την αξιολόγηση και το ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει και λογοδοσία. Όλα αυτά να τα εξισορροπούμε και με το ότι οι ε, φιλανθρωπικοί οργανισμοί ε, δουλεύουν προαιρετικά, δουλεύουν με μερική απασχόληση και δεν πρέπει να μετακυλήσουμε το διοικητικό άκτος σε αυτούς τους οργανισμούς. Ε, υπάρχει λοιπόν ε, ένα μεγάλο πεδίο όπου μπορούμε να συναντηθούμε. 517 είναι οι τροπολογίες που έχουν κατατεθεί. Είναι οι τροπολογίες από την Επιτροπή Γεωργίας, Περιφερειακής Ανάπτυξης, Προϋπολογισμών και ε, Γυναικών. Προσβλέπω λοιπόν στη συνεργασία με τους σκιώδεις και όλους τους εισηγητές έτσι ώστε να καταλήξουμε σε μια καλή πρόταση και να μπορέσουμε να συνεργαστούμε με ε, την Προεδρία. Και τέλος, κυρία Πρόεδρε, θέλω να σας πω ότι προτίθεμαι να συνεργαστώ στενά με την Ιρλανδική Προεδρία και ελπίζω να καταλήξουμε σε συμφωνία όσον αφορά στο πρόγραμμα αυτό. Ε, δεν έχουμε αρκετό χρόνο ε, στη συνάντηση του Απριλίου νομίζω ότι μπορούμε να επανέλθουμε και ε, μετά θα έχουμε παράλληλες συναντήσεις με το Συμβούλιο. Ευχαριστώ πολύ όλους σας και ε, προσβλέπω στις επόμενες εβδομάδες όπου πραγματικά θα έχουμε παραγωγική δουλειά. Ευχαριστώ. Αφήσετε ένα θέμα σχολίαστο. Την παρατήρηση της κυρίας Σρέτερ. θα ήθελα να το επαναφέρω, αν και δεν ήθεστε να σχολιάζει κανείς μετά τη δευτερολογία της συγγήτριας. Το πρόγραμμα αυτό βοήθησε τους απόρους. Γνωρίζουμε τι μάχη δώσαμε για να εγκριθεί και θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Να μην κατακαιρματίζουμε το θέμα της αλληλεγγύης και ο καθένας τον βολεύει. Το ίδιο, την ίδια συζήτηση είχαμε και για τη στρατηγική του 2020. Είπαμε αν θέλουμε και στόχο εκρίζωση της φτώχειας και αυτό το συζητήσαμε. Τελικά ελήφθη μια απόφαση και άσχετα με το σεβασμό των κανόνων της επικουρικότητας το αναγνωρίσα, αναγνωρίσαμε ότι και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης η άσκηση της αλληλεγγύης ε, προϋπέθεται κινητοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για την καταπολέμηση της φτώχειας. Οπότε αν θέλουμε να δώσουμε σάρκα και οστά στην ε, ιδέα της ελληνικής και μάλιστα εν μέσω μιας κρίσης όπου βλέπουμε όλοι ότι μη, ένας κρίκος της ε, αλυσίδας κρίσης είναι οι μακροοικονομικές ανισότητες μεταξύ των κρατών μελών και να λένε οι πλούσιες χώρες εμείς θα ασχοληθούμε με τους δικούς μας φτωχούς, οι υπόλοιποι να φροντίσουν τους δικούς τους. Προσοχή. Αν θέλουμε αλληλεγγύη, να τη φτάσουμε στα άκρα. Αλλιώς θα καταλήξουμε σε μια κατάσταση όπου εγώ εύπορος δεν έχω ανάγκη από εσά, βγάλτε τα πέρα μόνοι σας. Εντάξει, μπορεί να ε, υπερβάλλω κάπως, ε, αλλά προσοχή. Δεν θα πρέπει να αρκούμαστε σε μεγαλεπίβολα λόγια υπέρ της αλληλεγγύης και μετά να μην προβλέπουμε και έμπρακτη εφαρμογή της. Καλές οι φιλοσοφικές συζητήσεις, αλλά αν θέλουμε πραγματική αλληλεγγύη, θα πρέπει να είμαστε συνεπείς με τις προτάσεις μας και να εφαρμόσουμε την αλληλεγγύη προς όλες τις κατευθύνσεις, σε όλους και με δέσμευση όλων των κρατών μελών. Όχι επιλεκτική αλληλεγγύη. Ε, βλέπω ότι συμφωνεί η Ελίζα άρα όλα καλά. Όπως είπε και η καλά η συζήτηση άλλη φορά. Ολοκληρώνουμε λοιπόν αυτό το θέμα. Με ξεχνάτε ότι οι συμβαστικές τροπολογίες θα εξεταστούν στις 22 Απριλίου και θα τις ψηφίσουμε την ΕΠΑ αύριο, 23 Απριλίου. Θα πρέπει να τηρήσουμε αυτό το χρονοδιάγραμμα αν θέλουμε συζήτηση με την Ιρλανδική Προεδρία. Έχουμε και άλλα σημεία στην ημερήσια διάταξη, αλλά πιστεύω ότι θα διεκπαιρεώσουμε εντάχει. Σημείο 25. Ανταλλαγή απόψεως σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Όπως ξέρετε, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 7 η αρχική κρατών και 8 η Φεβρουαρίου, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων συμφώνησαν ε, ως προς τα ποσά, αλλά ε, κολυζέρισαν κάπως ε, ως προς τις νομοθετικές προτάσεις. Και ουσιαστικά με τα συμπεράσματά τους προδίκασαν κάποια θέματα της συναπόφασης. Η Συμφωνία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ε, προβλέπει έξι κεφάλαια στο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο με συγκεκριμένα ποσά που θα πρέπει να προσδιοριστούν ανάλογα με τις, οικονομικές, με τις νομικές βάσεις. Ό,τι αφορά το γενικό ανώτατο όριο μειώθηκε κατά 8% σε σχέση με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ό,τι αφορά τις θεσμεύσεις αναλύσεις υποχρεώσεων και μείωση κατά 9% σε ό,τι αφορά τις πιστώσεις πληρωμών του τέστην η αναλήψη υποχρεώσεων και οι πληρωμές με βάση την πρόταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν αποφάσισε να αμφισβητήσει αυτά τα ανώτατα όρια, οδηγούν σε προϋπολογισμό που αντιστοιχεί σε 1% της, ε, του κοινοτικού ΑΕΠ ε, για τις αναλήψεις υποχρεώσεων και 0,95% για τις πιστώσεις πληρωμών. Οπότε έχουμε ένα κοινοτικό προϋπολογισμό ε, που φτάνει στα όρια του προϋπολογισμού του 1987. Και πέραν ε, των σημείων που αναφέρθηκαν, έχουμε σοβαρές υπεφυλάξεις ε, σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα εκπλήρωση των πολιτικών στόχων, αλλά έχουμε πρόβλημα και με τα υπόλοιπα προσεκαθάριση, Τα ΡΑΛ που θα τεθούν στην Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων για το υπόλοιπο του φετινού προϋπολογισμού. Δεν χρειάζεται να σας υπενθυμίσω ότι είπαμε εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμα της προηγούμενης εβδομάδας. Απλώς να πω ότι για την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων διαπιστώσαμε κάποιες επιπτώσεις λόγω της πρότασης που αφορούν και την πρόταση ε, της πρωτοβουλίας για τους νέους ε, που προβλέπει χρηματοδότηση 6 δισεκατομμύριων ευρώ και την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την διατήρηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση και του Ταμείου για την ε, ενίσχυση των απόρων. Σε ό,τι αφορά τα μελλοντικά στάδια. Πέραν του ψηφίσματος ε, της περασμένης εβδομάδας, της 13ης Μαρτίου, θα πρέπει ε, να συμπεριλάβουμε τις επιπτώσεις των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις νομικές βάσεις που διαπραγματευόμαστε. Η βασική συνέπεια αφορά την ε, ανάληψη μιας πρωτοβουλίας υπέρ των νέων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τροποποίησε ήδη τις προτάσεις της, με βάση τις οποίες είχαμε εκπονήσει δική μας διαπραγματευτική εντολή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διόρθωσε δύο από τις προτάσεις της, στις 12 Μαρτίου. Αφενός την πρόταση για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, όπου πρόσθεσε μια αιτιολογική σκέψη, τροποποίησε τρία άρθρα, άρθρα και συμπεριέλαβε και την πρωτοβουλία για τους νέους και πρόσθεσε και ένα νέο κεφάλαιο με 8 άρθρα καθώς και ένα παράρτημα. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τροποποίησε την πρόταση κανονισμού CPR για το κανονισμό για τις κοινέ διατάξεις και πρόσθεσε μια νέα αιτιολογική σκέψη, τροποποίησε πέντε άρθρα, ένα παράρτημα και πρόσθεσε ένα ακόμη παράρτημα. Μετά από συζήτηση των συντονιστών, συμφωνήσαμε ε, να τροποποιήσουμε τη διαπραγματευτική εντολή για να λάβουμε υπόψη τις ε, αλλαγές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και η διαδικασία που αποφάσισαν οι πολιτικές ομάδες είναι η ακόλουθη. Οι συνάδελφοι μπορούν, στα αγγλικά δυστυχώς μόνο, γνωρίζετε πόσο μας πιέζει ο χρόνος, κατ' εξαίρεση εφαρμόζουμε αυτή τη διαδικασία. Οι συνάδελφοι λοιπόν μπορούν να υποβάλουν τις ε, ε, τροπολογίες τους στα αγγλικά μόνο μέχρι τις 25 Μαρτίου, Δευτέρα το μεσημέρι. Την επόμενη Δευτέρα το μεσημέρι δηλαδή. Εμείς θα προσπαθήσουμε να ε, τις εξετάσουμε, θα εξασφαλίσουμε κάποιο συντονισμό για να μπορέσουμε να συνυπογράψουμε πολλές τροπολογίες. Πάντως ο καθένας είναι ελεύθερος να καταθέσει τις δικές του. Στη συνέχεια ε, θα συνέλθουν οι διαπραγματευτικές ομάδες και των δύο κειμένων, ESF ε, του Κοινωνικού Ταμείου και CPR, με τους εισηγητές και σκιώδεις εισηγητές, την εβδομάδα ή την 15η εβδομάδα, στις αρχές της 16ης εβδομάδας, ε, για να καταλήξουμε στις συμβαστικές τροπολογίες και να εξασφαλίσουμε και μία συνάφεια των κειμένων, ώστε να μπορέσουμε να ψηφίσουμε στη συνεδρίασή μας στις 22ης και 23 η Απριλίου στην Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Οπότε θα τροποποιήσουμε τη διαπραγματευτική εντολή για το Κοινωνικό Ταμείο και ενδεχομένως θα τροποποιήσουμε και το κείμενο CPR. Επίση, απευθύνθηκα στον πρόεδρο της διάσκεψης των Προέδρων Επιτροπών, ζητώντας να κυρώσει την αποκλειστική μας αρμοδιότητα σε ό,τι αφορά την πρωτοβουλία για τους νέους. Αυτά ως προς το σημείο 25. Ενημερωτικά. Μήπως υπάρχουν παρατηρήσεις, έχετε απορίες. Όλα καλά. 250 τροπολογίες θα κατατεθούν για αυτά τα πέντε άρθρα. Όχι, ελπίζω. Περάμε στο επόμενο σημείο, το 26. Διαπραγματεύσει με το Συμβούλιο σχετικά με το πρόγραμμα για την κοινωνική αλλαγή και την καινοτομία. Το πρόγραμμα ΨΥ. Θα ήθελα να σας ενημερώσω με βάση το άρθρο 70 του κανονισμού για τα αποτελέσματα του τριμερούς διαλόγου που έλαβε χώρα στις 21 Φεβρουαρίου. Θα δώσω το λόγο στη Γιούτα Στάινρουκ για να μας ενημερώσει για την κατάσταση των διαπραγματεύσεων. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η, η τελευταία τριμερή συνάντηση ξεκίνησε 27 Φεβρουαρίου Ήταν η τελευταία συνάντηση με την Ιρλανδική Προεδρία ε, που σημαίνει ότι πρέπει κάπως να σημειώσουμε πρόοδο. Συμφωνήσαμε λοιπόν ότι στις, ε, στους τριμερείς αυτούς διαλόγους ε, θα συζητάμε περισσότερο με πολιτικές απόψεις. Η Προεδρία του Συμβουλίου συμφώνησε με αυτά που πρότεινε το Κοινοβούλιο. Κατ' ουσίαν πρόκειται για τις ε, συνοριακές συνεργασίες ε, υπό το πρόγραμμα OIRES. Στο μέλλον η χρηματοδότηση ε, θα παραμείνει υπό το πρόγραμμα της κοινωνικής αλλαγής και της καινοτομία, Η πρόταση της Κομισιόν ήταν όλα αυτά να χρηματοδοτηθούν από το Κοινωνικό Ταμείο οι συνεργασίες είναι διασφαλισμένες και με οικονομική συμμετοχή, όπως ακριβώς συνέβαινε και κατά το παρελθόν και νομίζω αυτό ήθελε και το Συμβούλιο, δηλαδή να υπάρξει συνέχεια. Όσον αφορά τώρα τις υπόλοιπες προτεραιότητες, Θέλω να σας πω ότι μέχρι τώρα δεν υπήρξε πρόοδος. Η επόμενη, ο επόμενος τριμερής διάλογος θα είναι στις 11 Απριλίου. Εμείς ε, εκ μέρους του Κοινοβουλίου Είμαστε σίγουροι ότι ε, δεν μπορούμε να περιστούμε σε αυτά που ε, μας έχουν υποσχεθεί μέχρι τώρα. Εμείς πιστεύουμε ότι έχουμε προετοιμαστεί πολύ καλά και ελπίζουμε το Συμβούλιο να το αναγνωρίσει αυτό. Και μόνο έτσι θεωρούμε ότι θα υπάρχει η δυνατότητα να έχουμε αίσιο τέλος στις διαπραγματεύσεις. Ευχαριστώ τον Σκιώδη Συγητή και τη Σκιώδη Συγητρία και την Πρόεδρο γιατί νομίζω ότι είμαστε μια πολύ καλή ομάδα ε, διαπραγματεύσεων. Ευχαριστώ πολύ και τη Γραμματεία. Πολύ ωραία. Θέλει κανείς το λόγο. Έχετε απορίες. Όχι, οπότε περνάμε στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, σημείο 27. χθες έλαβε χώρα ο 12ος τριμερής διάλογος Η γραμματεία ισχυρίζει ότι πρόκειται για τον ενδέκατο τριμερή διάλογο. Εγώ θεωρώ ότι είναι ο δωδέκατος, εν πάση περιπτώσει. Τους δέκα τριμερείς διαλόγους σίγουρα τους ξεπεράσαμε. Να δώσω το λόγο στην εισηγητριά μας, την κυρία Μωρά Σαχτιέ. Ευχαριστώ. Το θέμα δεν είναι πόσοι τριμερεί διάλογοι το θέμα, έγιναν, το θέμα είναι πόσο προχωρήσαμε στους τριμερεί διαλόγους. Το πρώτο σημείο που δημιούργησε μεγάλο πρόσκομα χθε με το Συμβούλιο αφορά ε, τις δύο ε, δικές μας παρατηρήσεις, το 25% για, ε, ε του Ταμείου Συνοχής που με βάση το κοινωνικό ταμείο αναφέρονται στο ε, ταμείο και το 20% του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου που προσημειώνεται για, το, για την καταπολέμηση της φτώχειας. Αυτά τα δύο ποσοστά, το 25% και το 20% που ε, τα κρατάμε για το ΕΚΤ και την καταπολέμηση της φτώχειας και αυτές οι δύο απαιτήσει ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν ικανοποιούν τα κράτη-μέλη και δεν είναι τις αρισκές του Συμβουλίου. Αυτό ήταν το θέμα του χθεσινού τριμερούς διαλόγου. Και με διάφορες τροπολογίες στο κείμενο αφισβητήθηκε το 25% του Ταμείου Συνοχής για το ΕΚΤ και το 20% για την καταπολέμηση της φτώχειας. Χθες όλα πήγαν ε, στραβά και ανάποδα. Δεύτερο θέμα, ο τίτλος του άρθρου 3. Ε, συζητήθηκε εκτενώς αυτό το θέμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βρίσκονται στο ίδιο, στο ίδιο μήκος κύματος ε, υπάρχει απόλυτη συμφωνία ώστε ο τίτλος να είναι πεδίο εφαρμογής, ενώ το Συμβούλιο θέλει να βάλει ως τίτλο προ... επενδυτικές προτεραιότητες, κάτι που δεν ανταποκρίνεται στο περιεχόμενο του άρθρου 3. Ζητήσαμε λοιπόν από το Συμβούλιο να μας πει ποια κρατημέλη ήταν υπέρα της α, αναφοράς αυτή στον τίτλο. Απάντηση όμως δεν λάβαμε. Και δεύτερο σημείο. Αυτός ο τίτλος ε, αν τροποποιηθεί, τι θα γίνει. Θα οδηγήσει στον διαχωρισμό του, σημείου, του άρθρου 3 σε, 3 δύο τμήματα, γιατί το πρώτο τμήμα μεν αφορά τις επενδυτικές προτεραιότητες, αλλά το δεύτερο τμήμα θα έπρεπε να περιλαμβάνει και μια διεύρυνση των επενδυτικών προτεραιότητων. Το Συμβούλιο λοιπόν θα πρέπει να διαβουλευτεί συντομότατα και πάλι με το Συμβούλιο για αυτό το σημείο. Τρίτο σημείο. Αρχίσαμε να συζητούμε το άρθρο 4 και Πέσαμε σε ένα σημείο απολύτως μη διαπραγματεύσιμο ε, δεδομένης της έκβασης ψηφοφορίας στην Επιτροπή μας. Το Συμβούλιο αυτό που επιθυμεί είναι να εισαγάγει την ιδέα ότι μπορούμε να καταλογίσουμε ως κοινωνική δαπάνη, δηλαδή σαν να προέρχεται από το ΕΚΤΕ, κονδύλια του ΦΕΝΤΕΡ, που έχουν κοινωνική χρησιμότητα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πώς εάν ε, φτιάξουμε ένα νοσοκομείο ή ένα βρεφονιπιακό σταθμό και αν χρηματοδοτηθεί αυτό από το ΦΕΝΤΕΡ για εξυπηρέτηση κοινωνικού στόχου, αυτό θα καταλογιστεί στο 20% του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε κάθετα αντίθετοι ε, με αυτήν την ιδέα και είναι πραγματικά σημείο ρήξης ε, για μας σας ε, μιλώ για το 25% του ποσοστό του ΕΚΤ, έτσι που κανονικά διοχετεύεται για την καταπολέμηση της ε, ένδυας. Είναι μη διαπραγματεύσιμο αυτό το σημείο, αλλά μπροστά μας έχουμε τείχο. Νομίζω ότι αυτό είναι ε, κέρια σημασίας. Κατόπιν, παράγραφος 4, παρά... εδάφιο 3. Οι προσθήκες που κάνουμε για να γίνει πιο ευέλικτος ο μηχανισμός ε, της θεματικής ομαδοποίησης που μας προτείνει το Συμβούλιο, κυρίως όταν μιλάμε για την κοινωνική καινοτομία και για την ε, ε, διασυνοριακή συνεργασία. Αυτά δεν θα συνυπολογίζονται όταν προσμετρούνται τα ε, ποσοστά και οι ελάχιστοι άξονε συγγνώμη, για την θεματική ομαδοποίηση. Για ποιο λόγο όλες αυτές ε, ε, οι παρακάμψεις του αρχικού κειμένου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με το οποίο είχαμε συμφωνήσει διότι λέει το Συμβούλιο πως πρέπει να καλυφθούν τα αιτήματα των μικρών κρατών μελών. Εμείς όταν βλέπουμε τις προσθήκες που έχει κάνει το Συμβούλιο και κάποιες τροπολογίες που κατατέθηκαν στη δική μας Επιτροπή συνειδητοποιούμε ότι δεν πρόκειται αποκλειστικά και μόνο για μικρά κράτη-μέλη ε, και τους ρώτησα πώς ορίζουν εκείνη τα μικρά κράτη-μέλη γιατί πόρο απέχουμε από, ε, ως προς τα συμπεράσματά μας ε, και φυσικά δεν διέφυγε της προσοχής μας αυτή η διαφορά. Εν κατακλείδη θα μπορούσα να πω πώς είτε πρόκειται για το 11ο ή το, το 11ο ή το 12ο Συμβούλιο, ε, ήταν κάκιστος αυτός ο τριμερής διάλογος, διότι είμαστε, ξαναλέω, στο χειρότερο σημείο Ρίξει ε, ω προς τα διαφορετικά οράματα που έχουμε από πλευρά Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Είμαστε στο ίδιο μήκο κύματο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματικά για αυτή την διαπραγμάτευση ε, και το Συμβούλιο είναι διαμετρικά αντίθετο. Σε τέτοιο σημείο που αναρωτιόμαστε αν ο απότερος στόχος του Συμβουλίου δεν είναι πραγματικά να θέσει σε κίνδυνο το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για την περιοδο 14-2014-2020. Ε, ε, έχουμε φτάσει στο ε, στο έσχατο σημείο από πλευρά τη Επιτροπής μας ως προς τις διαπραγματεύσεις και τις κινήσεις μπορεί να κάνει η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο. Ε, ίσως ε, θα πρέπει να ε, αλλάξουμε επίπεδο στις διαπραγματευτικές μας ομάδες, να ανέβουμε υψηλότερα και να ζητήσουμε τριμερή διάλογο με τους επιτρόπους. Λάσλο Άντορ και Γιωάννης Χάνε και τον Ιρλανδό, αρμόδιο Ιρλανδό Υπουργό, διότι οφείλουμε να διαπιστώσουμε ότι ε, δυσκολευόμαστε ιδιαιτέρως να ε, περάσουμε τη δική μας θεώρηση για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και πίσω από αυτά φυσικά το όραμά μας για την κοινωνική Ευρώπη ίσως ε, δεν κατάφερα καν να σας μεταδώσω την, το, βίο, το και κλίμα που επικρατεί στις διαπραγματεύσεις και την έντονη διαφωνία που υπάρχει. Ε, ο τέταρτ... Α, και να σας πω επίσης ότι στον πίνακα που χρησιμοποιούμε για τον τριμερή διάλογο το Συμβούλιο δεν συμπληρώνει ποτέ τη στήλη του. Ε, δεν έχουμε καν πληροφορίες για τη θέση του Συμβούλιου. Δεν είναι συμπληρωμένη η στήλη στον πίνακα. Ε, μάλλον ε, μεταχειρίζονται ελαφριά την καρδία αυτό τον τριμερή διάλογο από πλευράς ε, Συμβουλίου και Περιμένουμε μέχρι τις 12 το μεσημέρι τη Δευτέρα το να πω από τις ε, συζητήσεις του Συμβουλίου, ούτως ώστε να ξέρουμε ε, ε, τι μελγενέστε στις 27 στον επόμενο τριμερή διάλογο και 25 Μαρτίου τη Δευτέρα. Καταλαβαίνετε δεν μας αφήνει και αυτό πολύ χρόνο, δύο μέρες. Την Τετάρτη 27 προβλέπεται στις 6 η ώρα ο επόμενος ε, τριμερής ε, και στις 18 Απριλίου και 22 Απριλίου έπονται άλλοι δύο τριμερείς διάλογοι. Προσπάθησα, ε, Πρόεδρε, να αποτυπώσω πιστά τις χτεσινές συζητήσεις. Ο κύριος Σέρφης. Τρεις σύντομες παρατηρήσεις. Θα ήθελα πρώτα να επαναλάβω την αμέριστη υποστήριξη της σοσιαλιστικής ομάδας προς την ε, ε, κυρία Μωρά Σαρτιέ για όλο της το έργο, το προηγούμενο και το μελλοντικό. Είναι σημαντική αυτή η μάχη που δίνουμε για τη σωστή οριοθέτηση της ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής. Προσκρούμε απέναντι σε ένα τείχος, αυτό του Συμβουλίου, αλλά Όλοι οι τείχοι έχουν καταρρεύσει, ακόμη και οι τείχοι που υποτίθεται θα κρατούσαν μια ονειότητα. Γι' αυτό και σκόπιμο είναι να εκπονήσουμε μια ευφυή και αλληλέγγυα στρατηγική στο Ευρωπαϊκό, Συμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο επιτέλους να σταματήσει να επιδεικνύει τέτοια αυτιστική συμπεριφορά και να ακούσει και εμάς. Αν συνεχίσει το Συμβούλιο με τέτοια παιχνίδια τέτοια μικροτεχνάσματα θα χρειαστεί ε, να κάνουμε 20 και τριμερείς διαλόγους. Μας ενδιαφέρει να μάθουμε ποιες χώρες αντιστέκονται. Γιατί δεν χρειάζεται. Και εμείς ε, στόμα έχουμε και μπορούμε να μιλήσουμε. Ούτε κουφίμαστε, ούτε κουτσί. Θα πρέπει λοιπόν να μάθουμε ποιες είναι οι χώρες που αντιστέκονται και να προσπαθήσουμε να τις μεταπίσουμε. Θα πρέπει αυτέ οι συζητήσει να μην γίνονται κρυπτό και παραβίστο, αλλά μπροστά στα μάτια τη κοινή γνώμη. Ποιε είναι λοιπόν αυτέ οι χώρε, Φαίνεται ότι το Συμβούλιο εμπέζει πλήρω την κοινή γνώμη και την περιφρονεί. Γιατί αυτό δείχνει η περιφρονητική συμπεριφορά απέναντι μα. Γιατί δεν κατονομάζει τι χώρε, γιατί δεν εξασφαλίζει μια διαφάνεια. Έχει την πλήρη υποστήριξή μας, Ελίζαμπετ, είμαστε στο πλευρό σου. Το Συμβούλιο χρησιμοποιεί κάποιες τεχνικές ε, κολυσιεργίες και χρονοτριβείς. Εμείς θα προσπαθήσουμε να διασπάσουμε αυτή τη στρατηγική. Δεν μπορούμε να έχουμε τέσσερις υπαλλήλου από τέσσερις χώρες. Δεν ξέρω αν είναι και, μια, και ένα νησί αυτό που αντιστέκεται στο, στις προτάσεις μας για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Σας ευχαριστώ. Δεν βλέπω να υπάρχει κάποιος άλλος. Θα προσθέσω και εγώ δύο στοιχεία για το θέμα της διαπραγματευτικής τακτικής ε, του Συμβουλίου πρώτα απ' όλα, ε, διότι προσπαθήσαμε να ε, διακόψουμε, να αναχαιτήσουμε αυτή τη διαπραγματευτική πορεία χτες το βράδυ. Το είπε και η συγγήτριά μας, έχουμε ένα πίνακα με τέσσερι στήλες και στην τέταρτη στήλη δεν έχει τίποτα. Είναι άνευ προηγουμένου, έτσι, σε οποιοδήποτε τριμερή διάλογο και μετά από 12 τριμερείς διαλόγους παραμένει κενή η στήλη του ε, Συμβουλίου. Μένουμε άναυδοι. Δεύτερον, δεν ε, κατηγορώ κανέναν ε, ούτε τον πρώην εκπρόσωπο της Κυπριακής Προεδρίας ούτε και τον εκπρόσωπο της Ιρλανδικής Προεδρίας. Ούτως ή άλλως και στις δύο περιπτώσεις είχα εξαιρετικές σχέσεις με τους αρμοδίους υπουργούς και οι διαπραγματευτικές μας ομάδες ε, δυστυχώς δεν ήταν ε, στο επίπεδο των αρμοδίων υπουργών. Αυτό τι σημαίνει στην πράξη. Είναι ε, στρατηγικού χαρακτήρα οι διαπραγματευτικέ ε, τακτικέ, ναι, μεν, αλλά αντίκειται στην, ε, ε έννοια, στην αρχή τη συναπόφαση. Δηλαδή, τι γίνεται. Καταχωρούμε, καταλογίζουμε και τι κάνουμε, τα πετάμε μετά στις, στα σκουπίδια, δεν, δεν τα αξιοποιούμε. Δηλαδή, δεν υπάρχει επιστροφή, δεν διαπραγματευόμαστε, δίνουμε, υποχωρούμε, ξαναδίνουμε, ξαναδίνουμε. Και μία μέρα τι περιμένουμε να μας πούνε, ε, τι πρόκειται να γίνει, ποια είναι, τι διαπραγματευτική τακτική είναι αυτή, μας ε, θέτουν προτύχου, ε, έχουμε εξουθενωθεί όλοι μετά από 20 τριμερείς διαλόγους και τι λέμε, ή δεχόμαστε ή όχι τον Ιούλιο του 2013 για τα κονδύλια του 2014 μήπως πρέπει να περάσουμε στο επόμενο στάδιο αυτό προσπαθήσαμε να πετύχουμε χθε το βράδυ πρώτο στοιχείο, δεύτερο στοιχείο για την ε, διασύνδεση ανάμεσα στις διάφορες ε, διαπραγματεύσεις, ε, διότι το έκτε δεν είναι αυτόνομο, το μέλλον του είναι συνάρτηση της ύπαρξής του σε όλους τους υπόλοιπους τομείς και η ύπαρξη του σε όλους τους υπόλοιπους τομείς προσδιορίζεται από τις συνθήκες διαπραγματευτικές για, τις οποίες, για το CPR. Όμως ε, συνειδητοποιήσαμε ότι ήρθε η ώρα να κρούσουμε τον κίνδυνο του κινδύνου με μεγαλύτερη πυγμή ε, για το θέμα αυτό. Το άρθρο 84 είναι σημείο ρήξη. Εκεί μιλάμε για τις υποχρεώσεις ε, των κρατών μελών ε, ε, ανάλογα με το επίπεδο ανάπτυξη των περιφερειών σε σχέση με το ποιο ποσοστό της ε, πολιτικής συνοχής θα διοχετευτεί συγκεκριμένα στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και αναδιατυπώθηκε αυτό με τέτοιο τρόπο από το Συμβούλιο ώστε τα κράτη-μέλη δύνανται να καταργήσουν το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και τα, σας τα λέω αυτά και τα εννοώ. Πρέπει να... Ε, ε, ε, κρούσουμε με μεγαλύτερη πυγμή λοιπόν τον ε, κόδωνα του κινδύνου, τόσο ώστε στον επόμενο τριμερή διάλογο να εγείρουμε το πολιτικό ζήτημα με τη δέουσα σοβαρότητα. Στη δική μας Επιτροπή, οι ηθήνοντες των πολιτικών ομάδων παρακαλώ να το προσέξουν, διότι ε, στην Επιτροπή Απασχόληση και Κοινωνικών Υποθέσεων είναι τέτοιος ο ρόλος μας που πρέπει να εισακουστεί η φωνή μας. Όλοι αναγνωρίζουν πόσο σημαντική είναι η κοινωνική διάσταση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Όλοι αναγνωρίζουν τον κοινωνικό αντίκτυπο της κρίσης. Ε, μέσα στην έκθεση Tyson αυτά ψηφίσαμε. Ε, και όλοι ε, γαργαρίζουν μέσα στο στόμα τους όλα αυτά τα κοινωνικά ζητήματα. Ακόμη και οι κυβερνήσεις των κρατών μελών θέσπισαν το, τις για την νεολαία. Αν αφήσουμε όμως αυτό το άρθρο 84 του CPR όπως έχει τώρα, σήμερα, δεν θα υπάρξει στο μέλλον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ξεκάθαρο. Γι' αυτό το λόγο και ζητώ συγγνώμη που αργήσαμε ε, να ε, ξεκινήσουμε τις σημερινές μας εργασίες, αλλά μιλούσαμε με τον Επίτροπο Αντόρ. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε σε αυτό το στάδιο, κρίσιμο στάδιο της διαπραγμάτευσης. Λοιπόν, ε, είναι ε, κεντρική σημασία στο σημείο και ήθελα να επιστήσω την προσοχή σε αυτό. Ε, είναι πάρα πολύ καλό που συζητάμε για το στάδιο στο οποίο έχουν φτάσει πλέον οι διαπραγματεύσεις, γιατί πρέπει να ανασυνταχθούν οι διαπραγματευτικές μας ομάδες. Ε, τώρα φτάνω στο σημείο 28, τελευταίο σημασημερίσια διάταξη, σε πολύ σημαντική αντιπροσωπεία που πήγε στην, ε, στο Βερολίνο στις 13 με 15 Φεβρουαρίου. Ο Τόμας Μάνι ήταν εκεί, η κυρία Στάινμπρουκ, η κυρία Χάρκιν και εγώ. Τρία ήταν τα στάδια, στις 13 Ήμασταν στη Φραγκφούρτη, όπου κάναμε ανταλλαγές με τους ενδιαφερομένους για το ζήτημα των υπηρεσιών εδάφους. Οι υπηρεσίες εδάφους τους αερολιμένες ε, στα πλαίσια της έκθεσης ε, για την οποία γνωμοδότησε και η Επιτροπή μας ε, και η Επιτροπή Μεταφορών ε, απεφάνθη ε, επίσης και χθες. Κάναμε ανταλλαγή για την εταιρεία Manhaland που εντάσσεται και στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση διότι έλαβε βοήθειες και ε, ως συνήθως είναι όλα υποδειγματικά στη Γερμανία, οι κοινωνικοί εταίροι τα βρίσκουν μεταξύ τους και ούτω καθεξής και γι' αυτό διατηρείται το ταμείο δεύτερο στάδιο της ε, επίσκεψής μας στο Βερολίνο ανταλλαγή με τους βουλευτές της Μπούντεστα και της Υποεπιτροπής Μεταφορών συγκεκριμένα γι' αυτό ακριβώς το θέμα για τις ε, υπηρεσίες εδάφους στις 15 ανταλλαγή με την Υφυπουργό ε, του Υπουργείου ε, Κοινωνικών Υποθέσεων και Εργασίας. Ήταν εξαιρετικά πλούσια αυτή η ανταλλαγή απόψεων ε, και σχολιάσαμε πάρα πολλά ζητήματα. Πρώτα απ' όλα η Υπουργός, η μάλλον ε, επιχείρη για την απόφαση των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων για τη θέσπιση των εγγύσεων για την νεολαία και ανέπτυξε μια πλούσια επιχειρηματολογία βάσει της οποίας είναι ε, πάρα πολύ σημαντικό αυτό το σημείο τόσο ώστε να προωθήσουμε να προβάλλουμε την εικόνα της κοινωνικής Ευρώπης και να καταδείξουμε ε, αλληλεγγύη ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, για τις ε, εγγυήσεις αυτές εξέφρασε ε, και τις αμφιβολίες της η Υφυπουργός σε σχέση με το αν ενδείκνεται να διατηρηθεί το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση και το Ταμείο των Απόρων με επιχειρήματα που χοντρικά περιστρέφονται γύρω από την ικανότητα των κρατών μελών να καλύψουν τις δαπάνες που αυτό επισύρει. Βεβαίως, οι δυσκολίε των κρατών μελών ε, είναι συνάρτηση της ανάγκη διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας των κρατών μελών που δεν αντισταθμίζονται από την ύπαρξη ευρωπαϊκής βοήθειας. Ειλικρινά, εγώ το είπα και στην ε, Υφυπουργό ότι ε, ε, φάσκει και αντιφάσκει. Πώ υποστηρίζει από τη μια τι εγγυήσει για την νεολαία και από την άλλη δεν υποστηρίζει το Ταμείο Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση, το Ταμείο Βοήθεια για του Απόρου. Τώρα, για την κοινωνική εταιρική ευθύνη και τις ποσοστώσεις των γυναικών, καταλάβαμε ότι στην κυβέρνηση Μέρκελ αυτό το ζήτημα συζητείται πολύ. Ε, και δεν ε, υπάρχει απαραίτητα συμφωνία για όλα τα επιμέρους ε, σημεία. Αναφερθήκαμε επίσης στο θέμα της μεταβασιμότητας φορητότητας των συνταξιακών δικαιωμάτων και την συντάξιμων δικαιωμάτων και την απόσπαση των εργαζομένων. Η Υφυπουργό δήλωσε την αποφασιστικότητα που χαρακτηρίζει την γερμανική κυβέρνηση για τα βασικότερα σημεία της ε, διαπραγμάτευσης, άρθρα 9 και 12 συγκεκριμένα, πόσο σημαντικός είναι ο κατάλογος των κριτήριων που ε, δίνονται να ελέγξουν τα κρατη ή το πεδίο εφαρμογής της ε, κοινή και εξολοκληρου ολοκλήρου αστικής ευθύνης ήταν πάρα πολύ χρήσιμη και καρποφόρα η συζήτηση που κάναμε. Εν γέννη, ε, ειδικότερα η συζήτηση για την απόσπαση των εργαζομένων ε, ομολογουμένως ε, μας εξέπληξαν οι κοινωνικοί εταιροί γιατί βάσει πάγιας τακτικής της Επιτροπής μας συναντηθήκαμε ξεχωριστά με τους κοινωνικούς εταίρους στη Γερμανία, δεν ήθιστε όμως αυτό. Ε, και υπήρξε ένα μικρό προβληματάκι, ε, δυσκολία ερμηνείας από πλευράς τους, αλλά στη συνέχεια ε, το κατάλαβαν και δέχτηκαν ότι έτσι είναι οι του παιχνιδιού εδώ και αυτή είναι η πάγια τακτική της Επιτροπής μας και το δέχτηκαν. Χωρίς κανένα πρόβλημα, αυτά για την αντιπροσωπεία, ούτως ή άλλως γραπτός θα λάβει τα αναφορά για τις λεπτομέρειες όλων αυτών των διαβουλεύσεων.